So, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα τουλάχιστον σε όσους βρίσκονται εδώ. Πολύ. Σας παρακαλώ να καθίσετε. Και αφού καθίσετε, θα ήθελα μια και είναι περασμένες τρεις, να αρχίσουμε. Άρχεται λοιπόν και επίσημα η συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Περνάμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Τρεις αλλαγές έχω να προτείνω. Η πρώτη αφορά το σημείο 5. Ο συγητής δεν μπορούσε να έρθει σήμερα, γι' αυτό λοιπόν προτείνω το σημείο 5 της ημερησίας διάταξης να μετατεθεί για αύριο, 3η 14 Απριλίου στις 9 το πρωί. Εκεί δηλαδή όπου θα είχαμε το σημείο 8 για τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη. Ο συγητής της έκθεσης αυτής προτείνει να μεταφερθεί το σημείο αυτό στην επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει την 6η και την 7η Μαΐου. Και σημείο 20. Μηχανισμός επίλυσης εμπορικών διαφορών της Ένωσης. Για αυτό το σημείο θα ήθελα η συζήτηση να γίνει και κλεισμένων των θηρών. Τρεις λοιπόν αλλαγές στην ημερησία διάταξη. Υπάρχει κάτι άλλο. Ήδη το ανέφερε κύριε Πρόεδρε, για το σημείο 8 ήθελα να μιλήσω κι εγώ, να ζητήσω να παραταθεί, διότι δεν μπορεί να, να έρθει εδώ η συγγήτρια, διότι πρέπει να παρευρεθεί στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως ε, καλό είναι να αναβληθεί. Θα προλάβουμε το χρονοδιάγραμμα έτσι κι αλλιώς. Πολύ ωραία. Αν δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις, τότε θα εγκριθεί η μερίσια διάταξη όπως έχει τροποποιηθεί. Και λοιπόν το σημείο 5 θα συζητηθεί αύριο στις 9 το πρωί και το 8 στην επόμενη συνεδρίαση και το σημείο 20 θα συζητηθεί και κλεισμένον των θυρών. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έγκριση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης. Όπως συνήθως, εάν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης δεν έχουν διατυπωθεί σχόλια ή παρατηρήσεις, τότε θεωρούμε πως τα πρακτικά εγκρίνονται. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο σημείο 3, ανακοινώσεις του Προέδρου. Να σας υπενθυμίσω καταρχάς ότι αυτή η συζήτηση, αυτή η συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω web streaming σε όλο τον κόσμο. Είναι μια πολύ αγαπημένη μετάδοση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το κανάλι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ Δημοφιλέ λοιπόν μπορούν να μας δουν μέχρι και στη Νέα Ζηλανδία και να παρακολουθούν τις δραστηριότητες μας και από εκεί. Πήγαμε στο Ανόη του Βιετνάμ και στο Μίνχ ως αντιπροσωπεία. Επτά μέλη παρευρέθησαν εκεί από την αντιπροσωπεία και ο πρόεδρος. και δύο αντιπρόεδροι, ο κύριος Βίνκλερ, ο κύριος Ζαχραντήλ, ο οποίος είναι και ο εισηγητής ε, της έκθεσης για το Βιετνάμ, και οι δύο εκπρόσωποι του ΕΛΚ, ο κύριος Κασπάρη και από τους σοσιαλδημοκράτες ο κύριος Μάρτιν και η κυρία Ντεσαρνές, η κυρία Ροντρίγκε και ο κύριος Προύστ. Πιστεύω πως η αντιπροσωπεία βρέθηκε εκεί σε ένα πολύ σωστό χρονικό σημείο, κοντά στο τέλος των διαπραγματεύσεων και έτσι κατάφερε να αποκομίσει μια περιεκτική εικόνα της ε, κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις και μπόρεσε έτσι να ταυτοποιήσει πολλά προβληματικά σημεία. Συναντηθήκαμε με πολλούς υψηλόβαθμους εταίρους, μεταξύ άλλων τον Πρωθυπουργό του Βιετνάμ, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον αναπληρωτή Υπουργό Εμπορίου, τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ, προέδρους συνδικάτων και οικονομικούς εμπειρογνώμονες του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καθώς επίσης και εκπρόσωπους της κοινωνίας των πολιτών και της οικονομίας. Είχαμε λοιπόν πολλή δουλειά και πλούσιες εμπειρίες και πλούσια αποτελέσματα. Mm. Αυτό που κατέστη σαφές είναι ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον του Βιετνάμ για την οικονομική συμφωνία. Είναι μια προτεραιότητα για εκείνους Το TPP, για παράδειγμα, είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες για το Βιετνάμ. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να υποθέσουμε ότι το Βιετνάμ έχει και τη θέληση και την ετοιμότητα να ολοκληρώσει και να υπογράψει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Ιούνιο θα διεξαχθεί ο επόμενο γύρος των διαπραγματεύσεων και θα δούμε εάν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία τότε. Κάτι που θα αποτελεί μεγάλη επιτυχία και για τις δύο πλευρές, διότι το Βιετνάμ έχει μια μεγάλη, έχει ένα μεγάλο δυναμικό οικονομικό, το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Είχαν λοιπόν επιτυχία τα αποτελέσματα της ε, μετάβασης της αντιπροσωπείας μας εκεί και πιστεύω πόσο σημαντικές και χρήσιμες εμπειρίες. Μετά, όσον αφορά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την μακροοικονομική οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία, ψηφίσαμε στις 25 Μαρτίου με επιτυχία. Η έκθεση προήλθε από αυτήν εδώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο με διαβεβαιώνει ότι θα δρομολογηθεί η έκθεση. Επίσης, η ψηφοφορία για τα Δυτικά Βαλκάνια και για τις εισαγωγές υφασμάτων προβλέπεται στην Ολομέλεια της 29ης Απριλίου. έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επενδυτικούς φραγμούς. Η έκθεση αυτή παρουσιάστηκε το Μάρτιο και εντοπίστηκαν οι προβληματικοί τομείς στην Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία, την Αργεντινή και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Υπάρχει εκτενής αναφορά στις περιπτώσεις αυτές και στις χώρες αυτές. Πιστεύω πως αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Κατάινεν, ο οποίος είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, έχουν μεγάλο δυναμικό αυτή τη στιγμή. Και μπορούμε και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το δυναμικό. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μου. Υπάρχουν σχόλια. Κύριε Φινκλερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θέλω να θέσω ένα απλό ερώτημα διαδικαστικό. Δεν ξέρω αν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό αυτό που γίνεται σήμερα εδώ. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας κάτι, αλλά μήπως γίνει προηγούμενο δηλαδή ως μέλη της Επιτροπής εδώ δεν πρέπει να υποστηρίξουμε συγκεκριμένα συμφέροντα και αγορές. Εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις των ομάδων και των ομάδων συμφερόντων, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσουμε το προηγούμενο τέτοιου είδους διαφημίσεων να γίνονται δεκτές εδώ μέσα όπως αυτή που δείχνω. Και παρακαλώ το προσωπικό να ζητήσετε να αφαιρέσει τα αντικείμενα αυτά από την αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βίνκλερ. Ναι, αυτά τοποθετήθηκαν εδώ πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Φυσικά και υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες πως ε, θα διανέμονται μόνο αυτά που εγκρίνω σε κάθε συνεδρίαση και αυτοί οι κανόνες πρέπει να τηρούνται. Από ό,τι βλέπω προφανώς αυτά βρέθηκαν εδώ πριν την έναρξη της συνεδρίασης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν κάτι επίσημο που έχει πάρει την έγκριση αυτής της Επιτροπής. Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στο σημείο 4. Εμπόριο προϊόντων φώκιας. Η συγητής είναι ο κύριος Πέντσεν. Εδώ βρίσκεται. Πρόκειται για τροποποίηση της οδηγίας του 2009 Η οδηγία αυτή αφορά την απαγόρευση των προϊόντων αυτών τα οποία προέρχονται κυρίως από τον Καναδά και η οδηγία λοιπόν αυτή αφορά τα προϊόντα αυτά και τα οποία όπως είπα προέρχονται από τον Καναδά και από την κοινότητα των ε, Ινουιτών. Ο εισηγητή τώρα θα μας ενημερώσει για την κατάσταση και για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων και εδώ και με τον ΠΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα συνεχίσω στην μητρική μου. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δέχτηκαν έναν κανονισμό που απαγορεύει την πώληση παραγόγων προϊόντων φώκης στην Ευρώπη εναντίον αυτού διαμαρτυρήθηκαν ο Καναδάς και ο ΠΟΕ. Εγώ έχω τα εξή σχόλια για τους σκημόους, για τους Ινβίτ. Εγώ, έχουν προβλεφθεί ήδη δύο εξαιρέσεις παλαιότερα για αυτούς. Χωρίς να έχει αυτό όμως αρνητικές επιπτώσεις, χωρίς να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήματά τους. Αλλά το αποτέλεσμα τι ήταν. Δεν τους φερθήκαμε σωστά τελικά. Πολύ άδικα διότι Μερικοί κατοικούν σε πολύ απομακρυσμένα τμήματα του κόσμου και αντιμετωπίζουν δύσκολη κατάσταση. Αν χρησιμοποιούν τα προϊόντα φώκιας, χρησιμοποιούν τις φώκες για τρόφι, τα δέρματά τους για ρούχα κτλ. Επομένως αυτή η απαγόρευση καταστρέφει τον τρόπο ζωής τους. Η Κομισιόν μιλάει για τεχνικές προσαρμογής ώστε να μπορέσει να γίνει σεβαστή απόφαση του ΠΟΕ. Ξεχνάει όμως ότι η νομοθεσία που εγκρίνουμε έχει επιπτώσει στην καθημερινή ζωή ανθρώπων και δεν κατάλαβε, δεν έκανε, δεν ανέλαβε καμία σοβαρή μελέτη αξιολόγηση. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν εργάστηκε όπως έπρεπε. Εμείς θα ήθελαμε να κάνει την αξιολόγηση στα σοβαρά, γιατί οι αριθμοί που έχω εγώ δείχνουν ότι η νομοθεσία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή των Ινουίτ. Οι εξαγωγές δερμάτων φώκης έχουν μειωθεί κατά 400% περίπου, από 9 σε 2 εκατομμύρια τόνους. Εδώ μιλάμε λοιπόν για αυτόχθονες πληθυσμούς που έχουν την κακή τύχη να ζουν πολύ μακριά από τις Βρυξέλλες χωρίς σούπερ μάρκετ και μακριά και από τις συνήθεις εμπορικές ροές. Και έτσι εξαρτώνται από τη Γρυλανδία που αγοράζει αυτά τα δέρματα και επιχορηγεί και όλα στην πώληση αυτή, την αγορά αυτή. 135.000 ε, δέρματα φώκης έχουν αποθηκευτεί και σαπίζουν αυτή τη στιγμή στις αποθήκες. Θα έπρεπε λοιπόν η Κομισιόν, όπως λέει μια τροπολογία που θα καταθέσω, να λάβει υπόψη στην ειδική κατάσταση των Ινουίτες κοιμών και να δει πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσής τους ώστε να μην τους επηρεάζει αρνητικά η νομοθεσία που εγκρίνουμε. Πρέπει να γίνει λοιπόν μια βιώσιμη και σοβαρή αξιολόγηση για τους αυτόχθονες αυτούς πληθυσμούς που είναι και άνθρωποι που ζουν μαζί με τη φύση και συμπεριφέρονται πολύ φιλικότερα προς το περιβάλλον από εμά. Δεν τα έλαβαν αυτά υπόψη τους στις Βρυξέλλες. Η εξαίρεση τώρα για τη Βαλτική. Η Κομισιόν θεωρεί ότι πρόκειται για επίθεση, επίθεση, αλλά για κάτι πολιτικό δηλαδή, ενώ είναι τεχνικό το θέμα. Η εξαίρεση για τη Βαλτική αφορούσε ανέκαθεν έναν πολύ μικρό αριθμό φωκιών, φωκών και το θέμα εδώ είναι πώς θα σεβαστούμε περισσότερο το περιβάλλον. Αν καταργήσουμε την εξαίρεση αυτή τότε πάλι και εδώ θα παραμείνουν να σαπίζουν αχρησιμοποίητα και απούλητα δέρματα. Εμείς θεωρούμε τις φώκες ως πόρο, αυτό δεν έχει νόημα, η Κομισιό θεωρεί τις φώκες ως έναν απλό πόρο. Δεν είναι αυτός τρόπος βιώσιμης διαχείρισης όμως. Γι' αυτό προτείνω και μια άλλη αλλαγή. Εδώ γίνεται μια πολύ στενή ερμηνεία του κανονισμού. Θα ήθελα να συνεργαστεί μαζί μου η Κομισιόν για να δούμε πώς μπορεί να λυθεί το θέμα αυτό που δεν είναι μόνο τεχνικό αλλά και πολιτικό. Ο ατελής συμβιβασμό του 2009 θα μπορούσε και θα έπρεπε να διατηρηθεί. Το θέμα δεν είναι μόνο οι ποσοστώσεις και η κατανάλωση, υπάρχει και η οδηγία για για τα ενδιαιτήματα ή τους βιοτόπους, τους φυσικούς βιοτόπους. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέντσεν. Ο κύριος Λάιχτφριντ είναι σκιώδης εισηγητής για τους Σοσιαλδημοκράτε, αλλά ο κύριος Σούστερ ήθελε να τοποθετηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάιχτφριντ δεν είναι εδώ και μου ζήτησε να μιλήσω στη θέση του. Κυρίε και κύριοι, όπως γνωρίζετε, η απαγόρευση του εμπορίου προϊόντων φώκια έχει εγκριθεί από τον ΠΟΕ. Ζητείται μια βελτίωση των ε, τις οδηγίες και βελτίωση των εξαιρέσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Μπέντσεν για τη δουλειά που έχει κάνει στην έκθεση και ως κοιόδης εισηγητής των σοσιαλδημοκρατών θεωρώ πως ακολουθούμε μια μινιμαλιστική προσέγγιση και πως θα έπρεπε να είμαστε πιο πιστοί στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει ασκηθεί κριτική από τον ε, ΠΟΕ για τις ε, λεπτομέρειε του εμπορίου Φώκιας Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή στην εξέταση. Ορισμένες προτάσεις του εισηγητή χρειάζονται συζήτηση. Για παράδειγμα, η αίτηση για μια εκτίμηση αντικτύπου μετά από την απαγόρευση του εμπορίου στις κοινότητες αυτές που εμπορεύονται τα προϊόντα φώκιας. χρειάζεται ενδεχομένως να γίνουν κάποιες εξαιρέσεις για να προστατευτούν οι κοινωνίες αυτές. Και οι προτάσεις του εισηγητή για την βιώσιμη διαχείριση του εμπορίου μας βρίσκουν θετικά προσκύμενους. Φοβούμαστε ότι μία αναδιατύπωση θα οδηγήσει σε διακρίσεις Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε να, διαγρα... να μην διαγραφούν οι διατάξεις σχετικά με τις εξαιρέσεις. Σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με τον εισηγητή και θα χαρούμε για μελλοντικές συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάμπελ δεν είναι εδώ, ούτε κάποιος εκπρόσωπος των φιλελεύθερων. Υπάρχει κανείς από την ε, Γκουε, η κυρία Μουρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητής ε, προσπαθεί κάπως να ξεφύγει. Προσπαθεί να ε, δοθεί εκ νέου άδεια στο κυνήγι φώκιας ε, για τους αυτόχθονες ε, πληθυσμούς ε, που ζουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Δεν είμαστε κατά αυτών των παρεκκλήσεων, αλλά είμαστε κατά της εμπορικής προσέγγισης της όλης διαδικασίας. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου δεν θα δεχτεί αυτές τις τροποποιήσεις. Πρόκειται για παρεκκλήσεις οι οποίες δεν επαρκούν. Εάν δώσουμε αυτή τη δυνατότητα για τις παρεκκλήσεις, δεν θα υπάρχει δυνατότητα στη συνέχεια να αποφευθεί ε, η αλία μεγάλης κλίμακας. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να καταθέσουμε και σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος από τους πρασίνους, παρακαλώ. Θα συμφωνήσω και εγώ με την προλαλή σας και εμείς θεωρούμε ότι η έκθεση δεν μπορεί να ψηφιστεί ως έχει. Διαπιστώνουμε ότι μόνο ένα κράτος μέλος υπάρχει που μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτές ε, τις ε, ειδικέ ε, διατάξεις. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως μπορούμε να σβήσουμε αυτό το σημείο. Έπειτα, όσον αφορά τους Ινούιτες Κιμώους, αυτό που πρέπει να αποκλείσουμε είναι η εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων. Ούτε εδώ βρίσκουμε κάποιον λόγο να διαγραφεί αυτή η διάταξη όπως έχει προτείνει ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ και για την ομάδα EFTD. Και η κυρία Μπεγγίνε θα συμφωνήσω και εγώ με τους ε, συναδέλφους που έλαβαν το λόγο πριν από μένα και εμεί κατά την άποψή μας θεωρούμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί αυτό το οποίο έχει δεσμευτεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αφομιγή την αποφυγή εμπορίου παραγωγών προϊόντων φώκιας. Ε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ε, τα πιο περιζήτητα προϊόντα είναι των μικρών, μικρής ηλικίας ζώων που είναι από τριών ε, μηνών έως ενός έτους και η υπερθέρμανση του πλανήτη ε, θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση του συγκεκριμένου είδους. Επομένως ε, θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει η απαγόρευση των παραγωγών προϊόντων και θα πρέπει να προστατεύσουμε από αυτό το κυνήγι. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι αυτόχθονες πληθυσμοί επιβιώνουν από το κυνήγι φώκες, αλλά δεν είναι εύκολο να διακρίνουμε ποια ζώα προέρχονται από πρακτικές ε, που εφαρμόζουν αυτοί οι αυτόχθονες πληθυσμοί και ποια είναι προϊόντα ε, της όλης μεγαλύτερης επιχείρησης του κυνηγιού ε, φώκιας. Επομένως θα πρέπει να επαγρυπνούμε, να φροντίσουμε, να αποφύγουμε πολύ σημαντικές παρεκκλήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες μπορεί να είναι εις βάρος του συγκεκριμένου είδους και της επιβίωσής του. Επίσης θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο Καναδάς προσπάθησε να επιτεθεί στους κανόνες που ίσχυαν στο παρελθόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να ξέρω αν η ε, θέση σε ισχύ της συμφωνίας ΣΕΤΑ, δηλαδή της εμπορικής συμφωνίας με τον Καναδά, θα μπορούσε ίσως να θέσει ένα αμφιβόλο τη συγκεκριμένη νομοθεσία και να υπάρχει ο κίνδυνος ε, ο Καναδάς να μπορεί να επιβάλλει τροπολογίες ακριβώς λόγω της ε, συνθήκης αυτής ελευθέρων συναλλαγών. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο εκθεσής του, ε, τον κύριο Μπέντσεν. Όντω ε, πρόκειται για ακαθόδε ζήτημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σωστά. Αλλά το πιο σημαντικό, αυτό το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι να συμμορφούνται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με τι αποφάσει του ΠΟΕ. Το ερώτημα είναι πώ όμω, πώ θα το καταφέρουμε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Μπένσεν ε, πολύ σωστά λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το αντιμετωπίσουμε, η μέθοδος ε, που <laughs> προτείνει να υπάρξει συμμόρφωση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, είναι ε, λανθασμένη επιλογή, είναι μια πολύ κακή πρόταση να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε έτσι την νομοθεσία μας με τους κανόνες του ΠΟΕ. Θα πρέπει λοιπόν να τρέξουμε λίγο στο παρελθόν και να δούμε τι είπε η συγκεκριμένη επιτροπή όταν έγινε ε, δεκτή νομοθεσία. Εμείς κρούσαμε τον να του κινδύνου ακριβώς για να αποφευθεί αυτή η κατάσταση και στη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας είχαμε προτείνει να απορρίψουμε τη σχετική νομοθεσία. Και ο λόγος για τον οποίο προτάθηκε να απορρίψουμε την νομοθεσία ήταν γιατί εμεί ήμασταν τη άποψη ότι πρέπει το ζήτημα αυτό αυτή η βάναυση, παράλογη θανάτωση ε, φώκιας ε, ανά τον κόσμο θα πρέπει να καταδικάζεται, αλλά δεν θα πρέπει να λέμε ότι το εμπόριο αυτό καθ' αυτό είναι το πρόβλημα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπεσε ακριβώς την ίδια παγίδα και τώρα όπως και την πρώτη φορά. Είναι μια λύση η οποία θα είναι γρήγορη μεν, αλλά δεν θα είναι και η καλύτερη δυνατή επιλογή. Καταρχά, η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι οι νουίτ ε, του ε, Καναδά και τη Γρυλανδίας θα πρέπει να παίρνουν τι φώκες τους και να μπορούν να τις στέλνουν με τον κόσμο, αλλά οι φώκες οι οποίε ε, θηρεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν είναι με πιο ανθρώπινο τρόπο ε, από τον Ινουίτ θα πρέπει να απαγορεύεται. Αυτό θεωρώ ότι είναι κακή περιβαλλοντική πολιτική, κακή εμπορική πολιτική και είναι και ε, σαφής διάκριση. Ε, δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια εκτίμηση επιπτώσεων για να μπορέσει να ποσοτικοποιήσει τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής της πρότασης και αυτό αποτελεί ένα άλλο παράδειγμα μιας κακής λύσης σε μια κακή νομοθεσία. Τρίτον, θεωρώ ότι υπάρχει κάτι αντιφατικό. Δεν λέει απλώς ότι ε, επιτρέπεται κάποιος να θυρεύει φώκες, αλλά λέει ότι οι φώκες θα πρέπει να θυρεύονται για, σε μεγαλύτερο βαθμό λόγω της αύξησης του πληθυσμού τους. Ουσιαστικά ενθαρρύνει το κυνήγι φώκες, αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα προϊόντα της φώκες. Αυτό λοιπόν που θέλει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα είναι ότι συνεχίστε το κυνήγι, αλλά θεωρείτε ότι όλα τα παραπροϊόντα που παίρνετε είναι απόβλητα. Και αυτό δεν θεωρώ ότι είναι μόνο ε, άσχημα από δεντολογική σκοπιά, αλλά ε, παραβιάζει και την σύμβαση της βιοπικιλότητας από την οποία δεσμεύονται τα κράτη-μέλη. Λέμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε το κυνήγι φώκιας, αλλά μετά να τα καίμε τα προϊόντα και να θεωρούμε ότι είναι απόβλητα, διότι οι φώκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινδυνεύουν. Υπάρχει ε, αύξηση, ε, ραγδαία αύξηση του πληθυσμού. Αυτό είναι καλό, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι θα υπάρχει κυνήγη φώκιας και τώρα και στο παρελθόν. Το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε με τις ε, φώκες αυτές. Θα τις θεωρούμε απόβλητα, θα καίγονται, θα τις θάβουμε. Ε, ή θα χρησιμοποιούμε τις φώκες για να φτιάξουμε κάποια προϊόντα από ε, τα, τα ζώα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι η πρόταση δεν θα πρέπει να άρει την ε, εξαίρεση, αλλά να την τροποποιήσει, όπως πολύ σωστά προτείνει ο εισηγητής. Είναι πολύ σωστή κίνηση αυτή, διότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα και δεν προσπαθεί να δώσει μια σύντομη λύση. Να συνεχίσουμε το κυνήγι και να θεωρήσουμε τα προϊόντα είναι απόλυτα. Αυτό είναι άσχημη ε, περιβαλλοντική πολιτική, είναι κακή πολιτική και αυτό είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφεύγουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Ο κύριος Λάιφτφριτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που άργησα να γυρίσω, αλλά η Λουφτχάντζα ως ήθιστε καθυστέρησε σήμερα το πρωί. Στην αρχή δεν ήθελα να μιλήσω, αλλά μετά ο κύριος Φιέλνερ με οδήγησε στο να το κάνω. Εγώ έχω τελείω διαφορετική άποψη. Την τελευταία θητεία είχαμε νομοθετήσει καλά. Είχαμε ψηφίσει νομοθετήματα με μεγάλη πλειοψηφία. Όμως αυτή εδώ η περίπτωση είναι μια περίπτωση που δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιες αντιρρήσεις από την πλευρά του Καναδά. Αυτό που έχουμε αποφασίσει έχει ήδη αποφασιστεί και αυτό που πρέπει να φροντίσουμε είναι αυτά τα ζώα να μην σφαγιάζονται με αυτόν τον αποκρουστικό τρόπο που όλοι γνωρίζουμε. Και πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια των αποφάσεων του ΠΟΕ Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σωστή και δεν θεωρώ αναγκαίο να γίνουν πολλές αλλαγές. Είναι σχετικά σύντομη η πρόταση και πιστεύω πως είναι αρκετά καλή. Ευχαριστώ. Κύριε Φιέλνερ. Ίσως θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Θα ήθελα να πω το εξή στον κύριο Street. Καταρχά, δεν είναι μόνο η Lufthansa και άλλε εταιρείε ε, ε, έχουν τι ίδιε ε, περίεργε καθυστερήσει. Συμφωνώ όμω μαζί σα ότι το να προσπαθούμε να σταματήσουμε να σφαγιάζονται οι φώκες ε, ε, είναι λανθασμένο, αλλά εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποδείξετε γιατί εκφύσεως διότι ε, ουσιαστικά λέμε ότι οι Ινουίτ ποτέ δεν θα θανατάσουν με βάναυσο τρόπο τις φώκες, αλλά οι Ευρωπαίοι ε, κυνηγοί πάντα αυτό θα κάνουν. Γιατί αυτό ουσιαστικά περιγράφει συγκεκριμένη νομοθεσία. Λέει ότι δεν διορθώνουμε το πρόβλημα, αυτής της ε, αποτρόπαιας θανάτωσης των ζώων σε κάποιες περιοχές, λέμε ότι ως τη φώκια σκοτώσουν εννοείται εντάξει, ό,τι φώκια θανατάσουν οι Ευρωπαίοι πολίτε, ε, στους οποίους έχουμε την εξουσία και μπορούμε να νομοθετούμε, ε, θα επιτρέπεται. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση κάνετε λάθος. Voorzitter, ik ben blij te horen eh, πρόεδρε. Και ο κ. Φιέλνερ έχει προβλήματα με το θέμα του τρόπου της θανάτωσης των φωκών. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν ζητάμε χρήματα για την επιχορήγηση των προϊόντων αυτό δεν γίνεται δεκτό. Άρα πρέπει να θανατώνονται ακόμα περισσότερες φώκες. Αν επιτρέπεται το κυνήγι της φώκιας λόγω της εξαίρεσης για τους αυτόχθονες για να διατηρηθεί ο αριθμός του πληθυσμού δηλαδή αυτό πρέπει να είναι ο μόνος λόγος που δικαιολογείται εξαίρεση όχι εμπορικός λόγος να υπάρχει από τη στιγμή λοιπόν που ζητάμε χρήματα για τα παράγωγα προϊόντα φώκης ανοίγουμε το δρόμο στην γενικότερη εμπορία και εμπορική κατάχρηση. Ας πάμε ένα βήμα πίσω λοιπόν. Η Επιτροπή μας δεν γνωμοδότησε την προηγούμενη φορά για το θέμα των προϊόντων φώκης. Γιατί την προηγούμενη φορά δεν είχαμε μπορέσει να συνεδριάσουμε γιατί είχαν έρθει μέσα διαδηλωτές κλπ. Πρέπει να υπενθυμίσουμε όμως ότι πέρασε η νομοθεσία για τις φώκες με μεγάλη πλειοψηφία. Ο είπε ότι οι εμπορικοί περιορισμοί με θέμα, με δικαιολόγηση ευημερία των ζώων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Έγινε η συζήτηση για το κατά πόσον είναι ευαίσθητα όντα τα ζώα κλπ. Και τελικά εγώ δέχομαι την πρόταση, αυτή την πρόταση της Επιτροπής αυτή τη φορά και τα σχόλια του ΠΟΕ, αλλά αυτό που εννοεί ο κύριος Φιολνέρ είναι να παρεμποδιστεί η εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων φώκης και πρέπει να δείχνουμε μια συνέπεια στο διεθνές δίκαιο μέσα και έξω από την Ένωση. Ε, οι ίδιοι περιορισμοί πρέπει να ισχύουν. Αλλά είπαμε ότι η μόνη εξαίρεση είναι για λόγους ιστορικούς, πολιτιστικούς, οι Ινουίτ δηλαδή. Αν και ο ΠΟΕ μας είπε ότι δεν δικαιολογήσαμε όπως θα έπρεπε αυτή την εξαίρεση. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να γράψουμε, να συντάξουμε καλύτερα την διατύπωση της εξαίρεσης για τους εσκιμώους. Αυτό θα σταματούσε τους εμπορικούς κυνηγούς φώκης και μέσα και έξω από την Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάρτιν Λούκας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα θέλαμε και εμείς να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης και γιατί ε, συνεργάζεται μαζί μας για το έγγραφο αυτό. Θα ήθελα να υπενθυμίσω την απόφαση του ΠΟΕ, διότι από εκεί ξεκίνησαν όλα. Η απόφαση του ΠΟΕ θεωρεί ότι γενικότερα θα πρέπει να υπάρχει απαγόρευση για τα προϊόντα φώκια. Αυτό ήταν πολύ σημαντική λύση για την επίλυση αυτή τη διαφορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αναφέρθηκε και στι εξαιρέσει αυτή τη απαγόρευση. Η πρώτη εξαίρεση ήταν ε, για προϊόντα από την ε, διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και η δεύτερη εξαίρεση αφορούσε προϊόντα ε, κυνηγιού της κοινότητας των Ινουίτ. Όσον αφορά την ε, διαχείριση των θαλάσσιων αποθεμάτων, οπότε δεν δέχτηκε ότι αυτή η συμμορφή ε, ε είναι, αντίθετη, είναι διαφορετική από, την, από το κυνήγι που γίνεται στον Καναδά και στην Νορβηγία, επομένως αυτή η εξαίρεση αποτελούσε διάκριση. Το γεγονός ότι... Ε, το κυνήγι των Ινουάιτ ε, δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και είναι μικρή κλίμακα. Δεν θεωρούν ότι είναι επαρκέ επιχείρημα για να το διακρίνουν από τα όσα γίνονται στις άλλες περιοχές, στον Καναδά και στην Νορβηγία. Για τους Ινουίτ, ο ΠΟΕ δέχτηκε ότι το κυνήγι είναι διαφορετικό από το εμπορικό κυνήγι, διότι είναι απαραίτητο για αυτούς τους αυτόχθονες πληθυσμούς, για τους ε, σκημόους, ε, όπως αναγνωρίζεται και από το Διεθνές Δίκαιο και επομένω θα πρέπει να εξαιρείται από την απαγόρευση εμπορίας, διότι είναι απαραίτητο για την επιβίωσή τους, είναι απαραίτητο για την διαβίωσή τους να υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Πρόκειται για ουσιαστική ε, νίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το διασφαλίσει αυτό. Αυτό το οποίο είπε ο ΠΟΕ είπε ότι δεν ε, αναγνωρίζονται πουθενά θέματα ευημερία των ζώων σε αυτή την εξαίρεση ε, για τους Ινουίτ και δεν υπάρχει καμία σαφής διάκριση από την εμπορική δραστηριότητα. Αυτό λοιπόν ήταν αποτέλεσμα μετά από χρόνια διαμάχης η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπιζόταν με νύχια και με δόντια το κοινοτικό κεκτημένο και την απαγόρευση και τις απαγορεύσεις και τις απαγορεύσεις για τους θαλάσσιους πόρους, αλλά το αποτέλεσμα του ΠΟΕ είναι αυτό που είναι και πρέπει πλέον να τα αντιμετωπίσουμε. Εμείς έχουμε ακολουθήσει μια πολύ περιορισμένη προσέγγιση στην εφαρμογή βάση των όσων προβλέπει ο ΠΟΕ, όπως κάνουμε παραδοσιακά. Δεν είναι η πρώτη φορά που υποχρεούμαστε να αλλάξουμε νομοθεσία, ε, η τελευταία φορά που έγινε νομίζω ήταν πριν από 2-3 χρόνια όταν έπρεπε να αλλάξει ο κανονισμός για το του dumping μετά από την ε, αφισβήτηση από πλευρά Κίνας και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε την ίδια προσέγγιση. Δηλαδή, καταρχάς να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε στο ακέραιο το κεκτημένο, στο μέτρο του δυνατού και να γίνουν μόνο οι απαραίτητε αλλαγέ για να εφαρμοστεί η απόφαση του ΠΟΕ ταυτόχρονα η εφαρμογή να είναι αρκετά εύρωστη ώστε να ολοκληρωθεί η διαμάχη με τον ΠΟΕ και να αναγνωρίσουμε ότι η εφαρμογή αυτή είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει μία φορά, πρέπει να γίνει εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, πλαισίου ε, το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να θεώρησης από εκεί και πέρα της ε, διαδικασίας εφαρμογής. Ε, πρόκειται για μια προσέγγιση η οποία θεωρούμε ότι είναι δοκιμασμένη, είναι η ορθή προσέγγιση ε, στα όσα αποφασίζει ο ΠΟΕ για την εξαίρεση για τους αλάσσιους πόρους. Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να διασώσουμε αυτή την εξαίρεση αλλά η συνολική άποψη των νομικών επιρροχνωμόνων είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αν θέλουμε να εφαρμόσουμε στο κέρο αυτό που προβλέπει ο ΠΟΕ. Αν αλλάξουμε έστω και ελαφρά ε, τις προϋποθέσεις αυτής της εξαίρεσης, θα υπάρχει πάλι το πρόβλημα της διάκρισης ε, ε, για την εμπορική θύρα και θα πρέπει επίσης να δούμε ότι αυτό μπορεί να υποσκάψει την ίδια την διαδικασία. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση, μια περίπτωση τύπου κάτσε 22, όπου ε, το ίδιο το σύστημα έρχεται να ανατρέψει την ίδια την απόφαση. Τώρα, προτείνουμε λοιπόν να υπάρξει κάποια διατύπωση, η οποία θα αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ανησυχίες για την επιμερία των ζώων, στη συγκεκριμένη εξαίρεση και να υπάρχει μια ρήτρα ασφαλείας η οποία θα επιτρέπει να γίνεται διάκριση ε, από την εμπορική απαγόρευση. Και στόχος εδώ είναι να διατηρήσουμε μια ουσιαστική εξαίρεση για τους Ινουίτ που να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν οι Ινουίτ της Γρυλανδίας αλλά και αυτόχθονες πληθυσμοί αλλού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Και τώρα ο συντάκτης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος της παρέμβασής της, μιλώντας για το, τη σημασία της εξαίρεσης για τους Ινουίτ. Έχω ακούσει το ίδιο και από πολλούς άλλους σήμερα, γι' αυτό λοιπόν με χαρά άκουσα πως ζητείται μια εκτίμηση αντικτύπου του νομοθετήματος αυτού, έτσι ώστε να δούμε τις επιπτώσεις του στους ε, Ινουίτ της Γρυλανδίας. Και ελπίζω οι σκιώδεις ηγητέ να έχουν χρόνο για να διαβάσουν την μελέτη αυτή. Έχω μια μελέτη λοιπόν της ΒΒΕΦ. Μελέτη για τις εφόκες της Γρυλανδίας και το τι έχει συμβεί εκεί μετά τον κανονισμό. Και συμφωνώ με όσους είπαν σήμερα πώς πρέπει να διασφαλίσουμε ε, την ε, ανθρώπινη θανάτωση των ζώων αυτών. Όμως δεν είναι το ίδιο αυτό που κάνουν οι Ινουίτ και αυτό που κάνουν οι κυνηγοί για εμπορικούς σκοπούς. Οι νουίτ κυνηγούν φώκες για αιώνες τώρα και θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο βορρά του Καναδά γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν σε περίπτωση που απαγορευτεί το κυνήγι. Οι Ινουίτ σκοτώνουν τις φώκες και με το κρέας τους ε, τρέφονται οι ίδιοι, τα σκυλιά τους ντύνονται με τα δέρματά τους κλπ. Εδώ όμως υπάρχει και μία διαφορά ανάμεσα στο κυνήγι που κάνουν εκείνοι και στο κυνήγι για εμπορικούς σκοπούς όπου πάρα πολλά ζώα θανατώνονται και μάλιστα το χειμώνα όπου επικρατεί σκοτάδι όλο το 24ωρο. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω να συνεισφέρουμε με την έκθεσή μας σε μία λύση η οποία θα αντιμετωπίζει με υπεύθυνο τρόπο αυτές τις κοινότητες των Ινουίτ. Εδώ λέμε ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε μία απόφαση του ΠΟΕ. Υπάρχει νομοθεσία από τον Μάιο του 2014 Σχεδόν ένα χρόνο δηλαδή και τώρα ακούμε ότι θα επιβληθούν ποινές σε περίπτωση που δεν ακολουθήσουμε τις αποφάσεις. Τι κάνει η Κομισιόν με αυτό τον καιρό. δεν είναι μόνο οι τεχνικές προσαρμογές που χρειάζεται να γίνουν, πρέπει να γίνουν σεβαστοί και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κυνηγούν τις φώκες για να ζήσουν και δεν έχουν αρνητικές ε, επιπτώσεις οι πράξεις τους στο οικοσύστημα της περιοχής. Το θέμα λοιπόν είναι η βιωσιμότητα και όχι το εμπόριο. Το θέμα είναι η βιωσιμότητα μια ομάδα ανθρώπων ε, του οποίου ε, δεν έχουμε μεταχειριστεί και με τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω να βρούμε μια καλή για όλου λύση. Σα ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι η 17η Απριλίου στις 12 το μεσημέρι. Η έκθεση θα ψηφιστεί στην Επιτροπή στις 17 Μαΐου. Και μετά θα ψηφιστεί στην Αρμόδια Επιτροπή στις 14 Ιουνίου. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Όπως σας είπα το σημείο 5 έχει αναβληθεί για αύριο το πρωί. Τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών. Και σας περιμένω όλους εδώ μέχρι τις 4. Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε ξανά. Με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Κατάινεν. Καλώς ήρθατε. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην Επιτροπή μας. Και ελπίζω να συνεχίσουμε με έναν επικοδομητικό συνεχή διάλογο. Έχουμε πάρα πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Το θέμα των επενδύσεων και την τόνωσης της ανάπτυξης είναι μία από τις κυριότερες προτεραιότητες της εμπορικής πολιτικής. Και Είπατε ήδη πως είναι και μία από τις κύριες ε, δικές σας προτεραιότητες ε, το επενδυτικό σχέδιο και πως πρέπει να υπάρχει μία στενή συσχέτιση ανάμεσα στις επενδύσεις και στην εμπορική πολιτική. Έτσι ώστε αυτή η νέα αρχή για την Ευρώπη να μην έχει άσχημες επιπτώσεις για την ε, εμπορική πολιτική. Επίσης, σίγουρα θέλουμε να τονωθούν οι εξαγωγές και γι' αυτό δρομολογούνται σχετικές συμφωνίες, αλλά επίσης και να αυξηθούν οι συναλλαγές μας με τις τρίτες χώρες. Κάτι το οποίο θα συνεισφέρει πολύ θετικά στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Υπάρχει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη συσχέτιση ανάμεσα σε αυτά που κάνετε εσείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτά που κάνει η δική μας Επιτροπή. Σας καλωσορίζω λοιπόν ξανά και σας δίνω αυτή αμέσως το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων με μεγάλη μου χαρά και πανέτοιμος θα συζητήσω μαζί σας αυτά που μας απασχολούν από κοινού. Θα ήθελα όμως στην ομιλία μου να εστιάσω σε δύο από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το επενδυτικό σχέδιο και την ε, συμφωνία TTIP, την Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων. Και αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε να αποκομίσουμε πολύ μεγάλα ωφέλη εάν δρομολογηθούν ταυτόχρονα αυτές οι δύο συμφωνίες και εάν βρεθούν οι μεταξύ τους συνέργειες. Τον τελευταίο Νοέμβρη εγκρίναμε το επενδυτικό σχέδιο και τις προτάσεις για ρύθμις, τις ρυθμιστικές προτάσεις του EFSI, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει την εξέταση των προτάσεων και εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχουμε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σε εσάς. Και φυσικά ανυπομονούμε για τις επικοδομητικές συζητήσεις ανάμεσά μας και αναμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα το καλοκαίρι. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη νομοθετική πρωτοβουλία σε αυτήν την νέα κοινοβουλευτική περίοδο και πραγματικά όπως ε, συνηθίζουμε να λέμε, αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά, διότι στόχος μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Εάν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, πρέπει να ε, σταματήσουμε να εισαγάγουμε φραγμούς. Πρέπει να έρθουν λοιπόν αυτοί οι φραγμοί στο διασυνοριακό εμπόριο. Τους τελευταίους μήνες ταξίδεψα αρκετά στην ε, Ευρώπη προσπαθώντας να εξηγήσω το νέο επενδυτικό μας σχέδιο. Και αυτό που ακούω συχνά από εκπρόσωπους του ιδιωτικού τομέα είναι πως λείπει η, η πρόοδος στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και λείπει, λείπουν οι προσπάθειες για βελτίωση των επενδύσεων. Επίσης, στόχος μας θα πρέπει να είναι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν καλύτερη πρόσβαση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό έτσι ώστε να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε όσο περισσότερους πελάτες και να προστατεύεται η ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα. Η προσέγγιση αυτή ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου. Και πιστεύουμε πως, ε, όπως είπα και πριν, υπάρχουν πολλοί άλλοι λένε τομεί. Θέλουμε να προσελκύσουμε και εγχώριε επενδύσεις με τεχνογνωσία και νέο κεφάλαιο. Και αυτό σημαίνει πως πρέπει να δούμε τις ε, επιμέρους λεπτομέρειες και τις ε, κανονιστικές ρυθμίσεις διότι έτσι θα είμαστε σε καλύτερη θέση για να βελτιώσουμε τις ε, συνθήκες επιχειρηματικότητας ε, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, αν υπάρχει μια πραγματικά συνδεδεμένη ψηφιακή εσωτερική αγορά, τότε θα αυξηθεί η μόχλευση και η ισχύ μα στις ε, διεθνείς διαπραγματεύσεις. Επίσης, το επενδυτικό σχέδιο θα αυξήσει τα ωφέλη των της συμφωνία Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων στην εσωτερική αγορά και δημιουργώντας στρατηγικές επενδύσεις στον χώρο των υποδομών. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές στην παγκόσμια οικονομία. Το επενδυτικό σχέδιο έχει διατάξεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μελέτες που έχουμε κάνει μας δείχνουν συνέχεια ότι η έλλειψη κεφαλαίου είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων πέραν των σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να δοθούν κίνητρα και δυνατότητες στις μικρομεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις δυνατότητες που έχουν για επέκταση στο σε τις τρίτες χώρες. Προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε τους καλύτερους όρους για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και είμαστε σίγουροι πως και εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε τον ίδιο στόχο. Αυτή ε, τώρα η συμφωνία, η συμφωνία TTIP είναι μια τεράστια συμφωνία με πάρα πολύ μεγάλες ε, επιπτώσεις για όλους. Για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό διότι η συμφωνία αυτή είναι πολύ σημαντική για την ευρωπαϊκή οικονομία και θα αυξήσει την παρουσία μας στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα. Θα ήθελα να τονίσω ότι η ολοκλήρωση μιας τέτοιας συμφωνίας είναι εφικτή χωρίς να χαμηλώσουμε τα πρότυπά μας σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες, με την ασφάλεια των τροφίμων, με την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο πρόεδρος Γιούνκερ ο κύριος Αντιπρόεδρος Τίμερμανς και εγώ έχουμε συζητήσει με λεπτομέρειε την προσέγγιση μα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνεκτικότητα σε όλε τι ε, πτυχέ των διαπραγματεύσεων. Και η Επίτροπο ε, Μάλιμστρομ επίσης έχει δείξει την υποστήριξή τη ε, στο έργο μα. Έχουμε συζητήσει το πώ θα προχωρήσουμε σε σχέση με τι επενδύσει. και θα ήθελα να παραθέσω τα λόγια τη Επιτρόπου Μάλιμστρομ του τελευταίου μήνα. Μας είπε πως πιστεύει πως χρειάζεται ένα περιεκτικό κεφάλαιο για τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει ε, μη ε, ξεκάθαρες διτάξεις ε, που θα αφορούν μεταξύ άλλων και την επίλυση διαφορών επενδυτών κράτους. Όπως και η Επίτροπος Μάλιστον και εγώ ανυπομονώ να συζητήσω μαζί σας τους επόμενους μήνες πώς θα γίνουν αυτές οι αλλαγές, πώς θα προσελκύσουμε ξένο κεφάλαιο και πώς θα προστατεύσουμε τις επενδύσεις μας στο εξωτερικό ταυτόχρονα προστατεύοντας και το δικαίωμα των κρατών να έχουν ρυθμιστικό ρόλο. Προσπαθώντας λοιπόν να κάνουμε όλα αυτά, ελπίζω να διατηρήσουμε όλοι ανοιχτό μυαλό και να μην κλείσουμε πόρτες. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού υπάρχει μεγάλη, μεγάλο ενδιαφέρον στο τι γίνεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν με χαρά μου θα συζητήσω με εσάς και με όλους τους ε, ενδιαφερόμενους τις ε, λεπτομέρειες των ε, σχεδίων αυτών έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά ωφέλη και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους. Συμπερασματικά θα ήθελα να πω πως φέτος θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες και τις συνέργειες των μέσων που έχουμε στην εργαλειοθήκη μας για την βελτίωση της ανάπτυξης και την αύξηση των θέσεων απασχόλησης. Έχουμε την πρόθεση μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου να θέσουμε σε ισχύ ένα ε, νέο επενδυτικό σχέδιο, στο κέντρο του οποίου θα είναι η εξωτερική εμπορική πολιτική και το πώς θα καταφέρουμε να εξηγήσουμε με καλύτερο τρόπο το γιατί αυτές οι συμφωνίες θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης σε Ευρώπη. Κύριος στόχος μας λοιπόν είναι και η ενημέρωση των πολιτών με, διαφανό, με διαφανή τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν θα χαρούμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες μαζί σας. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ορισμένες προτεραιότητες στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου και φροντίζουμε να υπάρχει συνεκτικότητα. Χρειαζόμαστε όμως και τη δική σας στήριξη και συνεργασία. Κύριε Πρόεδρε, θα σταματήσω την ομιλία μου εδώ, ευχαριστώντας σας για την προσοχή σας και ελπίζοντας σε μια επικοδομητική συζήτηση και συνεργασία. Και όπως είπα, ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε της Κομισιόν. Θα δώσω το λόγο πρώτα στις πολιτικές ομάδες. Ο συντονιστής του ΕΛΚ που είναι κανείς δεν σηκώσει χέρι. Τότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Κλάικ από τους Σοσιαλιστάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Είπατε και εσείς αναφέρατε το TTIP είναι και για μας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Γιατί μιλήσαμε και με την κυρία Μάμστρομ και με τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων και αρχίζει να δημιουργείται η εντύπωση ότι όσο εμβαθύνεται τόσο γίνεται και πιο πολύπλοκη. Ποια νομίζετε ότι είναι τα κύρια προβλήματα που μπορεί να τεθούν στη διαπραγμάτευση, ας πούμε, οι γεωγραφικές ενδείξεις ή το άνοιγμα της αγοράς δημοσίων προμηθειών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέτοια πράγματα. Πώς το βλέπετε. Και δεύτερη ερώτηση, λίγο πιο στοχευμένη για το ISDS. Εδώ μέσα φαίνεται ότι γίνονται ενδιαφέρουσες και πολλές συζητήσεις για το θέμα. Οι σοσιαλιστές επιμένουν συχνά ότι η συνήθις μορφή του ISDS πρέπει να είναι αυτή που περιγράφεται και από την ΣΕΙΤΑ. Εσείς τι νομίζετε, διότι εγώ βλέπω ότι η παραδοσιακή μορφή του ISDS μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα. Μόλις μου ήρθαν οι τροπολογίες για την έκθεση ΛΑΝΚΕ περί TTIP και νομίζω ότι θα έχει πολλή δουλειά ο πρόεδρος 822 τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Θα μπορεί να βρεθεί λύση ή τι θα γίνει άμα δεν υπάρξει λύση. I would like to, to, to ask you. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σόλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Αντιπρόεδρε για την παρουσίασή σας. Πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα. Είχαμε και νωρίτερα στην Ολομέλεια, όχι στις Επιτροπές, συζητήσει το σχέδιο του Προέδρου της Κομισιόν για τις επενδύσεις. Κατά κάποιον τρόπο νομίζω ότι εδώ πρόκειται για βουντού, για μαγικά, διότι δεν κατάλαβα ακόμα και στη σημερινή ανταλλαγή απόψεων για τη διεθνές εμπόριο πώς είναι δυνατόν να ελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις να μας δώσουν λεφτά για αναπτυξιακά σχέδια ε, γιατί αν εξετάσω τα γερμανικά προγράμματα ας πούμε Πολλά από αυτά έχουν ήδη απορριφθεί εθνικώς ή επικρίνονται ε, εθνικώς ότι δεν αξίζουν τον κόπο, δεν θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, δεν έχουν νόημα για το βιομηχανικό μέλλον της Ένωσης ή της Γερμανίας αφού μιλάμε για τη Γερμανία. Αν λοιπόν μιλάμε για την βιομηχανία, για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και για την προώθηση πράγματι των επενδύσεων για να μην χαθεί η ορμή που είχε δημιουργηθεί μέχρι τώρα χωρίς να γνωρούμε βέβαια ότι περισσότερες, τα ε, περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έρχονται από την Κίνα πώς θεωρείτε ότι οι ε, επενδυτές θα μας δώσουν αυτά τα λεφτά. Τέλος, κάθε επένδυση πρέπει να ωφελεί, λένε, κάποια ιδιωτικά συμφέροντα, ιδίως μεγάλα, και κάποιο ρυθμό κέρδους. Ας πούμε, αν κατασκευάσουν γέφυρες ή δρόμους οι ιδιώτες επενδυτές, ο μόνος τρόπος να έχουν άμεσο κέρδος είναι με διόδια. Αν λοιπόν το αποτέλεσμα αυτής της επένδυσης είναι η αύξηση των διοδίων και η αύξηση των ιδιωτικών κερδών και των ιδιωτικών επενδυτικών προγραμμάτων, αεροδρόμια κλπ. Να μας το πείτε. Και αν αρχίσει ο κόσμος να χρησιμοποιεί εναλλακτικούς τρόπους, εναλλακτικούς δρόμους μάλλον, έξω των κυρίων αυτοκινητοδρόμων για να αποφύγει τα διόδια, τότε μπορεί το προβλεπόμενο κέρδος να είναι πολύ χαμηλότερο. Και τότε πώς θα αποπληρωθεί ο επενδυτής με δημόσιο χρήμα. Το δεύτερο θέμα, το TTIP, αναφέρθηκε. Και εσείς το αναφέρατε. Αν θελήσουμε να μιλήσουμε για την απασχόληση ή για την αγορά εργασίας, τότε δεν βλέπω τι πρόβλημα θα λυθεί. Μόλις επέστρεψα από τα Συνωμένα Πολιτείας όπου συνάντησα και συνδικαλιστάς στη Νέα Υόρκη και είναι και αυτοί, οι έχω αμφιβολίες για ως προς το κατά πόσον αυτές οι διαπραγματεύσεις θα φέρουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή την αύξηση των βελτίωση των συνθήκων εργασίας ή της απασχόλησης. Άρα η ανταγωνιστικότητα είναι ίσως κάτι επικίνδυνο αν θέλουμε να διατηρηθεί το κοινοτικό κεκτημένο στην Ένωση. Ή για την αύξηση, τη βελτίωση των αμερικανικών προτύπων στο επίπεδο των ευρωπαϊκών. Πώς μπορείτε λοιπόν να ελκύσετε επενδυτές από τη ΣΥΠΑ ας πούμε να έρθουν στην Ευρώπη και να επενδύσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Έχω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Εμπόριο. Βλέπουμε και στην έκθεσή σας ότι μας λέτε ότι το εμπόριο φέρνει αυτομάτως ανάπτυξη. Ιδιαίτερα στην όλη συζήτηση όμως για την TTIP υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δήλωση και ίσως θα μπορέσετε να μας διευκρινίσετε πώς πιστεύετε ότι θα συμβεί αυτό και ού μόνον αυτό πώς θεωρείτε ότι αυτό θα μας οδηγήσει και σε θέσεις απασχόλησης, διότι άλλωστε ήρθε και υπεύθυνο ε, επίτροπος για θέσεις απασχόλησης. Μπορεί ίσως να εξοικονομήσουμε κάποιες θέσεις εργασίας με τη συμφωνία, αλλά θα χάσουμε και θέσεις εργασίας και δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τον αριθμό των θέσεων που θα χαθούν. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς ε, ε, εξετάζετε καλύτερα την αγορά εργασίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς σκοπεύετε να δημιουργήσετε θέσεις εργασίας και ε, το εμπόριο δεν είναι το μόνο μέσο. Αυτό απειλεί και πολλές θέσει εργασία ανθρώπων που προσπαθούν να επιβιάσουν σε αυτόν τον κόσμο. Και επίσης μήπως θα πρέπει να εξετάσουμε και σε τοπικό επίπεδο τι αξία έχει δημιουργία θέσεων εργασίας και τι εσωτερική αξία πρέπει να δημιουργήσουμε με τις επενδύσεις που αναφέρατε. Βιώσιμες επενδύσεις για βιώσιμες θέσεις εργασίας και καλές θέσεις εργασίας. υποστηρίζουμε πάρα πολύ το γεγονός ότι ε, θα πρέπει να είναι κάτι βιώσιμο και εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι ακόμα βιώσιμη η όλη διαδικασία, διότι εξακολουθούμε να αυξάνουμε την ε, κατανάλωση σε ορυκτά καύσιμα και να μην ε, ε απλώς κατασκευάζουμε νέα οδικά δίκτυα. Αυτά δεν είναι επενδύσεις, είναι απλώς πατάλη χρημάτων. Επίσης, ε, τι θα γίνει με τις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής ε, ε, και το επενδυτικό σχέδιο, διότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή φαίνεται να αποκλείονται. Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια ώστε να πάνε εκεί που πραγματικά τα χρειάζονται. Και επίσης αναφερθήκατε και σε ιδιωτικές επενδύσεις. Στην Ευρώπη έχουμε ένα κενό επενδύσεων παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά κονδύλια διαθέσιμα, κυκλοφορεί χρήμα και κάποιοι προσπαθούν να δούνε πού μπορούν να επενδύσουν τα χρήματά τους. Ε, οι επενδύσεις όμως δεν υλοποιούνται. Και θα ήθελα να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντάξει, υπάρχουν όρια στο τι μπορείτε να κάνετε. Πού μπορείτε να πείτε ότι θα μπορούσατε να διοχετεύσετε πόρους για να επιληθεί το θέμα των επενδύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κίρτον Ντάρλινγκ. Θα ε, σταθώ σε κάτι διαφορετικό. Ε, θα συζητούμε την Τίτη όλο το απόγευμα. Εγώ θα ήθελα να ξέρω πώς το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό ε, Σχέδιο Επενδύσεων ε, ασχολείται με τη διεθνή διάσταση. σκοπεύουμε να κάνουμε κολοσιαίες επενδύσεις σε υποδομές και εξετάζοντας και τα προγράμματα τα οποία θα ε, χρηματοδοτηθούν θα υπάρξουν μεγάλα προγράμματα υποδομών που σημαίνει υλικά, ε, πρωτεσίλες ε, επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Αν εξετάσουμε την ε, κατάσταση ε, στις διεθνείς αγοράς, εγώ είμαι από την Βορειοανατολική Αγγλία και καταφέραμε να διασώσουμε την βασική μας επιχείρηση, την Plus ε, στη μέση της κρίσης και μας διέσωσε μια επιχείρηση από την Ταϊβάν, η SSI, η οποία έκανε επενδύσεις και ε, διέσωσαν την επιχείρηση αυτή η οποία κόντευε να χρεοκοπήσει. Και αυτή τη στιγμή οι επενδύσεις αυτές ε, ε κινδυνεύουν λόγω της τιμής ε, του χάλιβα παγκοσμίω και η κινέζικη οικονομία ουσιαστικά στέλνει τα πλεονάσματά της ε, στην παγκόσμια αγορά πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και όλες αυτές οι δυνατότητες που δημιουργούνται θα είναι προς όφελος και των βιομηχανιών μας και του εργατικού δυναμικού μας. Διότι αυτό αποτελεί βασική προτεραιότητα, θεωρώ, ε, για πολλού σε όλη την Ευρώπη, κυρίως σε περιοχές όπως τη δική μου, που είναι μία από τις φτωχότερε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ε, είναι αντίστοιχη με πολλές άλλες φτωχέ περιοχές της Ευρώπης. Υπάρχουν ε, βασικές βιομηχανίες συνήθως και αν αυτές οι βιομηχανίες κινδυνεύσουν από παγκοσμιοποιημένες αγορές, υπάρχει κίνδυνος για την τοπική οικονομία. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να συζητήσετε με την Επίτροπο Μάνστρα για να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτές τις διεθνές ε, επενδύσεις και πώς μπορούμε να προσφέρουμε ασφάλεια στους Ευρωπαίους εργαζομένους ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίσουμε ότι αντιμετωπίζονται καταλήλως και οι κίνδυνοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσει έχω. Η πρώτη έχει να κάνει με την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, η οποία ακύρωνε άλλες πρώτερες συμφωνίες και για τους Αμερικάνους ιδιαίτερα η συμφωνία TTIP είναι πάρα πολύ καλή διότι και δεν αποτελεί προβλήματα διότι έχουν άλλη νομοθεσία προστασίας των προϊόντων τους. Εμείς όμως δεν έχουμε αντίστοιχη νομοθεσία. Τι ε, θα κάνουμε σε αυτόν τον ε, τομέα, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. διότι σκεφτείτε και τις ε, τελευταίες αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Έπειτα, η δεύτερη ερώτηση που έχω να σας κάνω έχει να κάνει... Ή μάλλον όχι, θα μείνω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ στη μία ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχω και εγώ κάποιες πρόσθετες ερωτήσεις. Πιστεύω καταρχάς πως έχετε απόλυτο δίκιο ε, όταν μας λέτε ότι οι επενδύσεις είναι πολύ χαμηλές. Ακόμα και στη Γερμανία είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και αυτός ο κίνδυνος του να χάσουμε την ανταγωνιστικότητά μας προ όφελο κάποια άλλη τρίτη χώρα είναι υπαρκτό και πραγματικά χρειάζεται τόνωση τη ε, ανταγωνιστικότητα. Φυσικά, όμως, το πρόγραμμα έχει μόνο 300 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν είναι αρκετά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε στους περισσότερο νευραλγικούς τομείς έτσι ώστε να γίνουν στρατηγικές επενδύσεις. Για μένα ο πιο σημαντικός τομέας είναι η διαδικασία νέας εκβιομηχάνησης της Ευρώπης και το πόσο ψηφιακός ο κόσμος θα μπει στην διαδικασία παραγωγής. καθώς επίσης και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα πρέπει να υιοθετήσουμε. Και αυτά είναι κάποια μόνο, είναι τα κυριότερα από τα προβλήματα που έχουμε στον χώρο των επενδύσεων. Και αυτό με φέρνει στη δεύτερη ερώτηση που έχω να σας κάνω. Σε σύγκριση με τις Ηνωμένε Πολιτείε, εμείς δεν έχουμε μια παράδοση κεφαλαίου αντιμετώπισης κινδύνου. Ιδιαίτερα οι νέες εταιρείες όπως η Google για παράδειγμα ή η Amazon στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργήθηκαν με βάση αυτό το κεφάλαιο κινδύνου. Γι' αυτό λοιπόν παρατηρούμε ότι αυτά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα δημιουργούνται και ε, γεννιόνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι στην Ευρώπη. Πώς εσείς ε, βλέπετε την ικανότητά μας ε, για αυτά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Έπειτα, τρίτη ερώτηση, πόσο μπορούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια του ορίζοντα 2020 σε αυτό το σχέδιο επενδύσεων. Και εσείς μπορείτε να μας εγγυηθείτε το, πώς, το, το ότι θα γίνει με επιτυχία αυτή η σύνδεση Μπορείτε να μας δώσετε τις ίδιες εγγυήσεις εδώ όπως ε, για τον ορίζοντα 2020. Α, με συγχωρείτε, υπάρχει και κάποια... κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει να κάνει ερωτήσεις. Έχετε το λόγο, κύριε Μπόγκε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Προϋπολογισμού θα ασχοληθούν την επόμενη εβδομάδα με αυτό το σχέδιο επενδύσεων. Και θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να είναι κοινό μας στόχος να οδηγηθούμε σε ένα δίκαιο για όλους αποτέλεσμα. Ένα δίκαιο αποτέλεσμα καταρχάς για να στηρίξουμε αυτήν την πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Χρειάζεται να έχουμε αυτήν την αξιοπιστία. Είναι αναγκαία αυτή η αξιοπιστία για να διατηρήσουμε αυτό το πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να φροντίσουμε τόσο η δομή που θα έχουμε, η δομή των εργασιών μας, όσο και η χρηματοδότηση να ε, είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες και να έχουν την αναγκαία χρηματοδότηση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα από μέρους μου να παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι λίγο πιο δημιουργική από ό,τι υπήρξε στο παρελθόν σχετικά με την χρηματοδότηση προγραμμάτων. Είδαμε για παράδειγμα τη χρηματοδότηση του προγράμματος Γαλιλαίο και ε, είδαμε πως χρειάζεται περισσότερη ευελιξία και περισσότερη δημιουργικότητα και πως ακριβώς αυτά μας βοήθησαν να έρθουμε πιο γρήγορα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Όμως εγώ δεν άκουσα για τα σημαντικά επιμέρους ε, στοιχεία και τις λεπτομέρειες του, ε, του, πώς θα κάνουμε πιο εύκολη την, ε, το πιο εύκολο το έδαφος για επενδύσεις και πιο εύκολη την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε ακούσει για αυτά τα σχέδια ε, ανάκαμψης που ήταν ήδη από την προηγούμενη Επιτροπή Μπαρόζο, τα οποία θέλει να δραμολογήσει και η Επιτροπή Γιούνκερ, ιδιαίτερα στις χώρες που έχουν υποφέρει περισσότερο από τις τελευταίες ε, συγκυρίες. Όμως δεν αρκούν αυτά και δεν αρκεί μόνο η χρηματική υποστήριξη. Χρειάζεται ε, να δούμε και τι γίνεται στον ε, τομέα της ε, διοίκησης, της διοίκησης και του εμπορίου και το πώς θα ενισχυθούν αυτοί οι τομείς στα κράτη που παρουσιάζουν ελλείψεις. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως μας λείπουν αυτές οι προδιαγραφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα. Αυτό το βλέπω και στη δική μου εκλογική περιφέρεια. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε μια γέφυρα, που, ε, μια γέφυρα στη Βαλτική, έχουμε πάρα πολλούς ε, εμπλεκόμενους. Αυτή η γέφυρα, για παράδειγμα, στη Βαλτική θα συνδέσει τη Δανία με τη Γερμανία και θα ε, δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες και ε, στα δύο αυτά κράτη, αλλά και σε άλλα περισσότερα. Αλλά χρειάζεται πάρα πολύ καιρό. Ήδη πάνω από 10 χρόνια έχουν περάσει από τότε που είχαμε σκοπό να αρχίσουμε αυτή την κατασκευή. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα μόνο, κύριε Κατάινεν. Πώς λοιπόν θα δούμε τι θα βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις ε, λεπτομέρειες και τη διοικητική μας δομή έτσι ώστε να δώσουμε στις επενδύσεις ε, την ε, όθηση που χρειάζονται και έτσι ώστε να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε. Διότι, όπως σας είπα, δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση το πρόβλημα. Τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κατάινεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ομαδοποιήσω κάποιες ερωτήσεις. Οι πρώτε ήταν ερωτήσεις για την TTIP και μετά ρωτήσατε για το στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων. Για να σας δώσω λίγο το ιστορικό Η κυρία Κέλλερ μου είπε ότι φαίνεται να πιστεύω ότι το εμπόριο αυτομάτως ε, οδηγεί σε θέσεις εργασίας. Ε, λίγο πολύ πιστεύω το εξής. Παρά το γεγονός ότι εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρώπη, ξέρετε ότι είμαι Φιλανδός και πρόκειται για μία από τις χώρες όπου ο ρόλος του δημοσίου του τομέα είναι ε, πολύ ε, υψηλός, ίσως και λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε αλλά προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η χώρα θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ε, στους πολίτες της και παιδεία υψηλού επίπεδου, η χώρα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική στον κόσμο, αν όχι και η πιο ανταγωνιστική στον κόσμο, προκειμένου να μπορεί να ε, κάνει εμπόριο και επιτυχώς. Διότι μόνο μέσω εμπορίου μπορεί η χώρα να χρηματοδοτεί ε, το κράτος πρόνοιας. Αυτό λοιπόν είναι το υπόβαθρο. Γι' αυτό και εγώ υποστηρίζω ακράδαντα την εσωτερική αγορά. Εάν δεν πίστευα ε, στο εμπόριο θα άρχιζα να δημιουργώ φραγμούς ε, με τα κράτη-μέλη και ε, να μειώνεται η ενιαία αγορά σε τομείς ο οποίους είναι αναπτυγμένοι. Θεωρώ ότι πιστεύει ότι χρειαζόμαστε μια αγορά στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τις υπόλοιπες περιοχές της Ευρώπης και αυτή είναι η λογική που διέπει τα πάντα. Η κυρία Κέρτον Ντάρλινγκ μας έδωσε ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς μπορούν να πάνε στραβά τα πράγματα όταν δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες. Ε, υπάρχουν καλές επενδύσεις ε, στη Χαλιβουργία και αν δεν υπάρχουν καλοί κανόνες εμπορίου, κάποιες άλλες χώρες είτε θα κάνουν dumping είτε θα επιδοτούν ε, την ε, ίδια τη βιομηχανία που δημιουργεί προβλήματα ε, πιο συγκεκριμένα στην περιοχή σας, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για να υπάρχει λοιπόν μια βιώσιμη λογική επένδυση, εάν μάλλον υπάρχει μια βιώσιμη λογική επένδυση και υπάρχει μια τέτοια πολιτική, μπορεί να γίνει άχρηστη. Πρέπει λοιπόν να επενδύουμε σε πράγματα τα οποία δεν θα επιτρέπουν στους ανταγωνιστές μας να χρησιμοποιούν αθέμητους τρόπους ανταγωνισμού και με αυτόν τον τρόπο να καταστρέφουν τις θέσεις εργασίας μας εδώ στην Ευρώπη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία αναφερθήκατε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πάρα πολύ προσεκτικά τα πράγματα προκειμένου να διαπιστώσει αν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε θέματα εμπορίου. στις διαπραγματεύσεις για την τύπη αρχίζουμε να μπαίνουμε στα πιο δύσκολα ζητήματα και όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Λάικτριτ, αυτά είναι τα πιο ακαθόδη. Αν εξετάσουμε όμως ε, την κατάσταση αποθετικής σκοπιάς, ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε επιτύχει με κάποια πράγματα, αλλά έχουν παραμείνει όλες οι δυσκολίες αυτή τη στιγμή. Όπως είπε και ο πρέσβης, ο κύριος Φρόμαντ στη... Ε, στο τραπέζι Ε, του Ομπάμα ε, λέει ότι υπάρχουν τα δύσκολα πράγματα θα είναι πάντα δύσκολα. Επομένως, εάν θέλουμε να έχουμε μια δίκαιη συμφωνία εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ σκληρά και να σταματήσουμε να κατηγορούμε τους Αμερικανούς και να λέμε ότι δεν είναι σοβαροί με το τάδε ή οι Ευρωπαίοι δεν είναι σοβαροί με το δίνα. Αυτό μας οδηγεί σε αδιέξοδο. Υπάρχουν μια σειρά από πολύ δύσκολα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το θέμα των κρατικών προμηθειών για τους Αμερικανούς που επιθυμούμε εμείς και υπάρχουν πράγματα που επιθυμούν οι ίδιοι και είναι πολύ διαφιλονικούμενα για μας. Εάν όμως υπάρξει ισχυρή δέσμευση, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ μας. Από πολιτική σκοπιά αυτό είναι πάντα πολύ δύσκολο, αλλά ούτως ή άλλως γι' αυτό γίνονται οι διαπραγματεύσεις, για την επίλυση των δύσκολων θεμάτων, γιατί τα εύκολα έχουν ήδη επιληθεί. Τώρα, το σύστημα επίλυσης διαφορών, το ISDS, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό τμήμα της συμφωνίας. Ε, γνωρίζω όλες τις επικρίσεις, οι οποίες εν μέρη ε, έχουν κάποια σημασία, εν μέρη όμως οφείλονται σε πολλές παρανοήσεις και πρέπει να σας μιλήσω ανοιχτά. Ε, λογικά υπάρχουν ανησυχίες και όσον αφορά το σύστημα επίλυσης διαφορών, τουλάχιστον για μένα και για ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το θέμα δεν είναι άσπρο μαύρο, δεν είναι ή καλό ή κακό. Έχουμε μια αξιολόγηση και βάσει αυτής χρειαζόμαστε το ISDS προκειμένου να προστατεύουμε τις επενδύσεις. Διότι αν η νομοθεσία των ΗΠΑ δεν επιτρέπει ίσα δικαιώματα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όπως στις αμερικανικές επιχειρήσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά προκειμένου να υπάρξει μια δίκαιη μεταχείριση ε, από το δικαστικό ε, σύστημα των Αμερικανών. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέραν αυτού όμως υπάρχουν και κάποιες ε, θεμελιώδεις αξίες ε, από, και από τις δύο πλευρές και τουλάχιστον εμείς από πλευράς Ευρώπης θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ε, τα κοινοβούλια ή οι χώρες θα έχουν δικαίωμα προσφυγής και να τα ρυθμίσουν αυτά τα πράγματα. Σαφώς θα είναι σημαντικό το ζήτημα αυτό στο μέλλον. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα όσον αφορά την TTIP είναι και το γεγονός ότι ακόμα υπάρχουν κάποιες θεμελιώδεις αξίες τις οποίες πρέπει να προασπίσουμε. Αλλά αυτό είναι τμήμα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Μεταξύ αυτών πρέπει να ρυθμίσουμε και αυτό. Να περάσω τώρα στο στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων. Όπως θα γνωρίζετε, το σχέδιο επενδύσεων έχει τρία τμήματα. Το πρώτο, και αυτό το οποίο έχει συζητηθεί περισσότερο, είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, αυτό το νέο ταμείο. Το δεύτερο τμήμα είναι ε, τα ε, έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν μαζί με αυτό το συμβουλευτικό κόμβο και το τρίτο είναι η ρύθμιση της νέα αγοράς. Εγώ θα επικεντρωθώ κυρίως στο ταμείο τώρα και θα πω και δύο λόγια για τα έργα. Ο κύριος Σόλτς ρώτησε πώς μπορούμε να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις. Και η κυρία Κέλλερ ρώτησε για ποιο λόγο ε, καθυστερούμε σε επενδύσεις. Υπήρξαν και κάποιες ερωτήσεις ε, για το πώς θα μπορούσαν να επωφεληθούν οι πλέον ευάλωτες χώρες από τα κονδύλια του Ταμείου. Πρώτον, το νέο ταμείο δεν θα αποτελεί πανάκια. Πρόκειται για ένα ταμείο το οποίο είναι επικεντρωμένο σε συγκεκριμένα πράγματα υπό την έννοια ότι επικεντρώνεται στις ιδιωτικές επενδύσεις και σε κάποιες περιπτώσεις σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Δεν θα δανείσει χρήματα σε ε, αμυγός ε, δημόσιες επενδύσεις. Επίσης, Πρόκειται για ένα ταμείο το οποίο είναι επικεντρωμένο σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα γιατί επικεντρώνονται σε προγράμματα υψηλότερου κινδύνου. Προγράμματα τα οποία δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τη συνήθι δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ιδάλλως ε, ε, θα μπορούσαμε να κεφαλαιοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την αφήνουμε να δανείζει περισσότερα ε, στα προγράμματα που δανείζει ούτως ή άλλως. Ε, πέρσι δάνεισε περίπου 77 δις και σε αιτήσια βάση ε, σε, μεταξύ 60 και 70 δισεκατομμυρίων οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεις. Τώρα, το νέο ταμείο, το οποίο θα είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα επικεντρωθεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να προσελκύσουμε ιδιωτικού πόρους, διότι ο ιδιωτικό τομέα μας λέει ότι υπάρχει ρευστό, δεν μας λείπει το ρευστό, αυτό που μας λείπει είναι χρηματοδότηση ε, η οποία να, να επιμερίζει τον κίνδυνο. Και αυτό θα προσπαθήσει να καθορίσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ε, εν μέρη θα μοιράζεται τον κίνδυνο των ιδιωτικών επενδυτών στα έργα τα οποία είναι τόσο επικίνδυνα ή μάλλον πιο επικίνδυνα από άλλα. Είναι τόσο επικίνδυνα που ο ιδιωτικός τομέας από μόνος του δεν θα μπορούσε να αναλάβει το βάρος του κινδύνου. Παραδείγματο χάρη, ρωτήσατε πώ μπορούν να υποφαληθούν οι πιο ευάλωτε χώρε από αυτό. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ε, παρέχει αυτό το στοιχείο ε, επιμερισμού κινδύνου και περιλαμβάνει και τον κίνδυνο τη κάθε χώρα. Προσφάτω επισκέφτηκα την Κύπρο και μου είπαν ότι χρειάζεται μια επένδυση μικρού μεγέθους στον τουριστικό τομέα. Παραδείγματος χάρη, ανακαίνιση ξενοδοχείων, ε, του συστήματος υδροδότησης, των αγωγών υδροδότησης, πρόκειται για μικρής κλίμακας επενδύσεις. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, ο εκάστοτε ιδιοκτήτης, είναι διατεθειμένος να επενδύσει στο ξενοδοχείο του, αλλά επειδή υπάρχει ο κίνδυνος της συγκεκριμένη χώρας, το ε, χρηματικό κόστος είναι αρκετά υψηλό η συμβουλή μας ήταν η εξής. Γιατί να μην βρείτε διάφορες επενδύσεις και να υπάρχουν κάποια στοιχεία επιμερισμού κινδύνου ε, μέσω του EFSI, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και έτσι το κόστος χρηματοδότησης για τον ε, επιχειρηματία θα μειωθεί και θα μπορεί να ανακαινιστεί το κάθε ξενοδοχείο και να μπορέσουν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους ή να ε, δουλεύουν την επιχείρησή τους μακροπρόθεσμα. Αυτό λοιπόν κάνει το Ταμείο. Επικεντρώνεται σε προγράμματα υψηλότερου κινδύνου, τα οποία ε, δεν μπορεί να αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας από μόνος του. Ένα δεύτερο στοιχείο, το οποίο σχετίζεται πολύ ε, στενά και με το θέμα το οποίο έθεσε κάποιος συνάδελφος, εάν δανώσουμε χρήματα και δώσουμε κεφάλαιο κινδύνου σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο φαίνεται να συζητείται ευρύτερα όπου ε, πήγα και στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ε, ε, κάνουν έρευνα και ανάπτυξη θα μπορούσαν ίσως να λάβουν και πιστώσεις από τράπεζες, τουλάχιστον στη χώρα μέλος τους κάθε φορά, αλλά δεν μπορούν να λάβουν δανειοδότηση γιατί δεν έχουν ένα αντίκρισμα να, δώσουν. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Και αν βοηθήσει το Ταμείο θα μπορούσαμε να έχουμε πελάτες και στη Γερμανία και τις κάτω χώρες και στην Κύπρο και αλλού. Εμέσως δηλαδή θα χρηματοδοτούμε έρευνα και επενδύσεις, έρευνα και ανάπτυξη και φυσικά αυτό ε, σε συνδυασμό με την πραγματική οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Ο λόγος ε, για τον οποίο δεν υπάρχουν επενδύσεις ε, δεν είναι ένας, υπάρχουν αρκετοί. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει ζήτηση. Δεύτερον, κάποιες χώρες σε κάποιους τομείς δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικές παγκοσμίω. Τρίτον, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει έλλειψη ρευστού, υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης στην οποία υπάρχει και επιμερισμός κινδύνου. Και όπως σας είπα και μόλι προηγουμένω, το γεγονό ότι δεν υπάρχει ε, αντίκρισμα είναι πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν θέλουν να ζητήσουν δανειοδότηση. Ε, και ε, φυσικά και η σταθερότητα της περιοχής είναι ένας τομέας ο οποίος ε, επηρεάζει τις επενδύσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα φάσμα μέτρων, το οποίο περιλαμβάνει και λύσεις σε εθνικό επίπεδο, σε ανταγωνιστικότητα. Χρειαζόμαστε και ευρωπαϊκά εργαλεία, τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν ώστε να υπάρξει καταμερισμός του κινδύνου και επίσης θα πρέπει να δημιουργήσουμε και ε, ε, νέες αγορές. Και γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντική και η νέα αγορά, διότι όπως γνωρίζουμε όλοι, από τα κεφάλαια, για παράδειγμα, από τα παραδείγματα που έχουμε στη ψηφιακά προϊόντα. Αν προσπαθεί κάποιος να αγοράσει ψηφιακά προϊόντα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι και παράνομο. Ε, κυρίως στον ψηφιακό τομέα και στο δεσυνοριακό εμπόριο. Στον ενεργειακό τομέα επίσης δεν υπάρχει πλήρως εναρμονισμένη εσωτερική αγορά. Γι' αυτό ακριβώ χρειάζεται βελτίωση των νέων αυτών αγορών. Ορίζοντας 2020. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικότερα ζητήματα. Όταν θα ξεκινήσουν οι τριμερείς διάλογοι σίγουρα θα βρεθεί μια λύση, αλλά να σας εξηγήσω λίγο τη λογική που υφέρπει. Ο ορίζοντας 2020 είναι το μεγαλύτερο επενδυτικό ε, ταμείο, ταμείο ε, έρευνας. Είναι 50% μεγαλύτερο από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε 3,5% που σημαίνει 2,7 δις τα χρήματα αυτά θα χρηματοδοτηθούν ως ε, χρηματοδοτικό μέσο, δηλαδή ως μέσο μόχλευσης για να υπάρξουν επενδύσεις, για παράδειγμα, για τον τομέα της έρευνας. Βέβαια, πολλοί τώρα λένε ότι η έρευνα δεν μπορεί να επωφεληθεί από τα χρηματοδοτικά μέσα. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι ε, θα πρέπει να καταβληθούν και οι μισθοί των καθηγητών και των διδασκόντων από το δημόσιο τομέα. Αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι και ο ε, ιδιωτικό τομέα χρειάζεται επενδύσεις. Ε, μόλις πήγα στην Γαλλία και στην Κύπρο, όπως σας είπα, και μας είπαν με ιδιαίτερη περηφάνεια τι επενδύσεις έκαναν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βοήθησε ιδιαίτερα σε κάποια πανεπιστήμια και υπήρξαν επενδύσεις σε έρευνα. Επίσης, αρκετά πανεπιστήμια μας είπαν ότι σκοπεύουν με τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσουν σε εγκαταστάσεις έρευνα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει καθημερινά και πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις και στην έρευνα και αυτό ε, γίνεται εν μέρη με τον ιδιωτικό τομέα, κυρίως όμως με τη βοήθεια ε, του δημοσίου τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν αυτά τα 2,7 δις θα χρησιμοποιηθούν ως πίστοση ή ε, για να προσελκύσουν πολύ περισσότερα κονδύλια από τα χρηματοδοτικά μέσα. Μια τελευταία παρατήρηση για το θέμα αυτό. Αν εξετάσετε τις χώρες τις οποίες η έρευνα και η ανάπτυξη ε, έχει μεγαλύτερη αναλογία ε, στο ΑΕΠ. Σε εκείνες τις χώρες υπάρχουν και επιδοτήσεις αλλά πολλά χρηματοδοτικά μέσα επίσης. Η πραγματικότητα λοιπόν δεν είναι ασπριμαύρη. Καταλαβαίνω ότι πρέπει κάπως να καταβάλλονται μισθοί. Αυτό ισχύει και θα ισχύει και για το μέλλον. Αλλά ε, εάν επενδύουμε σε δικές εγκαταστάσεις ε, χρειαζόμαστε και χρηματοπιστωτικά μέσα. Ελπίζω Α, ε, κάτι επιπλέον, διότι αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που από ό,τι φαίνεται δημιουργεί κάποιες παρανοήσεις το Σεπτέμβριο το Συμβούλιο Κοφίν αποφάσισε να δώσει έναν ενδεικτικό κατάλογο δυνητικών επενδύσεων. Ο λεγόμενος κατάλογος της Task Force έτσι έγινε γνωστός και δημιουργήθηκε εξή παρανόηση ότι όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο κατάλογο θα χρηματοδοτηθούν είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φαίνεται ότι κάποιοι θεωρούν ότι η χρηματοδότηση για τα συγκεκριμένα προγράμματα ε, είναι ε, ε, με μορφή πιστέσεων. Από όσα σας είπα τίποτα δεν ισχύει. Ο κατάλογος δεν έχει άμεση σχέση με το σχέδιο επενδύσεων. Είναι μάλλον ένας ενδεικτικός κατάλογος. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά προγράμματα. Υπάρχουν πολύ καλά διαρθρωμένα επενδυτικά προγράμματα του δημοσίου τομέα, αλλά επειδή ακριβώς είναι αμυγός δημόσια, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από αυτά τα κεφάλαια κινδύνου. Υπάρχουν πολύ καλά έργα του ιδιωτικού τομέα, δυστυχώς πολύ λίγα και αν αυτό ο οποίος προωθεί το ιδιωτικό πρόγραμμα ε, ενδιαφέρεται όντως σοβαρά, μπορεί να αποτανθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και να ρωτήσει ε, αν είναι κατάλληλο για χρηματοδότηση ή αν θα μπορούσε να πάρει χρηματοδότηση ε, με τη συνήθεια εδώ μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι σαν μια τράπεζα στην οποία οι πελάτες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα οι κυβερνήσεις δεν επιλέγουν τα προγράμματα, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιλέγουν. Επαφίεται στον ιδιωτικό τομέα ή σε αυτές τις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα να υποβάλουν την αίτησή τους και να δουν αν υπάρχουν και πόροι και ίσως θα μπορέσουν να υπάρχουν και κάποια ε, στοιχεία επιμερισμού κινδύνου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε μου. Αυτό ήταν βέβαια μία απλή αρχή του διαλόγου μας για την προώθηση των επενδύσεων της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Good, liebe Μάλιστα. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 7. Το αγαπημένο μας θέμα τελευταία, η TTIP. Σήμερα έχουμε σκοπό να συζητήσουμε τις τροπολογίες, τις οποίες λάβαμε στο σχέδιο έκθεσης η προθεσμία ήταν η 26 Μαρτίου. Και στο μεταξύ της μέτρησα 898 τροπολογίες υποβλήθηκαν. Αυτό λοιπόν σημαίνει πως χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο έτσι ώστε να μεταφραστούν όλες οι τροπολογίες σε όλες τις γλώσσες. Δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες ακόμα. Με μεγάλη προσοχή λοιπόν κοίταξα αυτές τις 898 τροπολογίες και θα προσπαθήσω τώρα να δω πώς θα καταφέρουμε να οδηγηθούμε σε έναν ε, συμβιβασμό με, το να ενώσουμε ορισμένες από αυτές. Και μετά από αυτήν την αρχική ενδελεχή εξέταση πρέπει να πω πως βλέπω πως η γενικότερη κατεύθυνση των ε, τροπολογιών και του σχεδίου έκθεσης. Είναι λίγο πολύ ίδια. Ορισμένες φορές υπάρχουν καλύτερες διατυπώσεις ή αναδιατυπώσεις, αλλά σε γενικές γραμμές πηγαίνουμε όλοι στην ε, ίδια κατεύθυνση και πιστεύω πως δεν θα έχουμε επομένως ε, δυσκολίες να φτάσουμε σε έναν επικοδομητικό συμβιβασμό. Και είμαι απόλυτα πεπιτισμένος ως εισηγητής πως θα καταφέρουμε να δώσουμε την κατάλληλη ακρίβεια χωρίς να χαθούμε στις λεπτομέρειες και χωρίς να θυσιάσουμε αυτήν την ακρίβεια στο βωμό των πολιτικών μας πεπιθήσεων. Μετά λοιπόν από αυτή την πρώτη εξέταση μπορώ να διαπιστώσω πως υπάρχουν τέσσερις ε, κάπως αμφιλεγόμενοι τομείς. Ο πρώτος είναι ο τομέας της προστασίας των δεδομένων, όπου παρατηρώ διαφορετικές απόψεις που φαίνονται στις τροπολογίες. σχετικά με τις ε, προϋποθέσεις ε, της προστασίας δεδομένων. Δεύτερος τομέας είναι η παροχή υπηρεσιών και αυτό είναι ένα θέμα που χρήζει μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις μεθόδους δηλαδή που θα ακολουθηθούν. Ο τρίτος τομέας είναι ο τομέας της ευβιωσιμότητας, το συγκεκριμένο κεφάλαιο λοιπόν, για τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και Επίσης, όπως κατέστη σαφές, ε, τόσο ζήτημα για την επίλυση διαφορών επενδυτή κράτους. Αυτοί λοιπόν είναι οι τέσσερις ε, τομείς τους οποίους υπάρχουν οι περισσότερες διαφωνίες, οι περισσότερο αμφιλεγόμενοι τομείς και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια κοινή λύση. Ε, Καταρχάς, Είχαμε δεχτεί γνωμοδοτήσεις από πολλές επιτροπές, 14 στον αριθμό. Επτά επιτροπές ήδη μας κατέθεσαν τις ε, γνωμοδοτήσεις τους. 16 Απριλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία, την πέμπτη δηλαδή, οπότε μέχρι τότε θα έχουμε λάβει και τις υπόλοιπες 7 ε, γνωμοδοτήσεις και θα συγκεντρώσουμε όλη την εμπειρογνωμοσύνη των επιτροπών αυτών στη δική μας έκθεση. Ακριβώς λοιπόν εξαιτίας αυτού του τεράστιου αριθμού των ε, τροπολογιών και του μεγάλου αριθμού των γνωμοδοτήσεων από τις άλλες επιτροπές, Συζήτησα με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και με τους συντονιστές και ζήτησα να δώσουμε κάπως μια παράταση στις προθεσμίες. Εισακούστηκε αυτή η παράκληση μου λοιπόν και θα ψηφίσουμε την έκθεση όχι στις, ε, στις αρχές Μαΐου όπως ε, είχε προβληθεί, αλλά στις 28 Μαΐου. Έχουμε λοιπόν δύο εβδομάδες παραπάνω χρόνο για να συζητήσουμε και εάν γίνει αυτό, θα πάει έκθεση στην Ολομέλεια προς ψήφιση τον Ιούνιο, τη δεύτερη εβδομάδα αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν θα έχουμε εμείς εδώ την δυνατότητα, κάτι που είχα ζητήσει κιόλας από την αρχή, να έχουμε μία ισχυρή πλειοψηφία για τις τροπολογίες και για την έκθεση στο σύνολό της. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα να έχουμε μία ισχυρή πλειοψηφία στην ψηφοφορία, διότι σίγουρα θέλουμε να τοποθετηθούμε απέναντι στην θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό θα το καταφέρουμε όχι με μια πολύ μικρή πλειοψηφία, αλλά με μια πολύ ισχυρή πλειοψηφία. Έτσι θα δώσουμε και, μια, και ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Και είμαι επίσης πεπισμένος ότι χρειαζόμαστε αυτήν την πολύ ισχυρή πλειοψηφία έτσι ώστε να κάνουμε την θέση μας απόλυτα σαφή προς τις Ηνωμένε Πολιτείες. Και δεν σας κρύβω ότι έχω κάποιες ανησυχίες. Και ο αντιπρόεδρος Κατάινεν μας είπε πριν από λίγο ότι χρειάζονται φιλοδοξίες και από τις δύο πλευρές. Και είμαι σίγουρος πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτήν την φιλοδοξία που χρειάζεται. Αυτό φάνηκε και στις διαπραγματεύσεις εξάλλου. Οι προτάσεις τους όμως δεν ήταν για εμάς φιλόδοξες. Και χρειάζεται να παρακολουθούμε και τις εξελίξεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο για να δούμε την προθυμία που δείχνουν εκεί για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και βλέπουμε πως υπάρχουν μεγάλες επιφυλάξεις και πως είναι διχασμένο το Κογκρέσο. Δεν είναι καθόλου γνωστό το πώς θα ψηφίσει το Κογκρέσο. Και από την άλλη παρατηρούμε ότι στις Ηνωμένε Πολιτείε προτεραιότητα δεν είναι η TTIP αλλά η αντίστοιχη συμφωνία για τον ειρηνικό. Και μετά την ολοκλήρωση εκείνης της συμφωνίας θα δείξουν περισσότερη φιλοδοξία απέναντι στην συμφωνία ΤΙΤΙΠ. Γι' αυτό λοιπόν θα επιθυμούσα και εμείς να δώσουμε ένα ξεκάθαρο στίγμα για το τι ακριβώς θέλουμε και να δείξουμε και την δυναμική μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Για να μπορέσουμε όμως να το κάνουμε αυτό, όπως είπα, χρειάζεται μια ισχυρή πλειοψηφία. Βρισκόμαστε πριν από τον 10ο κύκλο των διαπραγματεύσεων για την Συμφωνία TTIP και όπως είπα και πριν, δεν βλέπω ότι έχουμε χρησιμοποιήσει στο έπακρο όλο το δυναμικό μας. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα αρχικά εισαγωγικά λοιπόν. σχόλια από εμένα. Το λόγο έχουν τώρα οι σκιώδεις εισηγητές, αν είναι εδώ. Και μετά το λόγο έχουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι αυτής της Επιτροπής. Η κυρία Ρόβαλτ κυρία Πεκλάκη επίσης, αλλά νομίζω πως έχουμε εδώ την κυρία Σάκε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχηθώ καταρχάς καλή τύχη. Νομίζω πως είστε αρκετά θετικός και αρκετά φιλόδοξος. Θα ήθελα λίγο να σταθώ στην ουσία των τροπολογιών τις οποίες υπέβαλα, οι οποίες πιστεύω πως αντανακλούν και τις υπόλοιπες ε, τροπολογίες και το σκεπτικό των τροπολογιών της ομάδας μου των ε, φιλελευθέρων. Η συμφωνία TTIP θα έχει πολύ σημαντικές ε, επιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα η φιλοδοξία μας. Και πρέπει να φροντίσουμε να πιέσουμε από τη μία τους διαπραγματευτές μας, αλλά και να τους εξοπλίσουμε. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε όλοι μαζί έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μία συμφωνία TTIP η οποία θα δώσει όχι μόνο ωφέλη στις επιχειρήσεις αλλά θα ανοίξει και νέους δρόμους για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέα πρόσβαση, κάτι που είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό ως εφηλελεύθεροι. Χρειάζεται να αρθούν οι φραγμοί ταυτόχρονα διατηρώντας τα πρότυπα τα οποία έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνοντας υπόψη επίσης και τις νέες εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας. Υπάρχει η κοινή δήλωση για τις ε, δημόσιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεωρώ αρκετά θετική και που αναφέρεται σε πολλούς για μας σημαντικούς τομείς όπως η πρόσβαση στην αγορά. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε το πόσο επίγουσα χρονικά είναι η πρόοδος αυτών των ε, διαπραγματεύσεων. Διότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα, ιδιαίτερα στην ε, ασφάλεια των ε, τροφίμων. Οι δικές μας τροπολογίες επίσης εστιάζουν στη, στον παγκόσμιο αντίκτυπο της Συμφωνίας TTIP και στο πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να διατηρήσει την ποιότητα ζωής που έχει και να μην ε, επιδεινωθούν μέσω της συμφωνίας αυτές οι συνθήκες ζωής, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τις επόμενες γενιές. Θεωρούμε πως πρέπει να δοθεί έμφαση στις ε, νέες τεχνικές, ε, στις νέες τεχνολογίες, στους νέους ε, τρόπους εμπορίου. Είμαστε εστιασμένοι στο μέλλον. Ο αντίκτυπος επίσης του ψηφίσματος θα πρέπει να αντανακλά και τις εξελίξεις στο παγκόσμιο γίγδεστε. Δεν είναι φυσικά το τελικό ψήφισμα και το τελευταίο ψήφισμα σχετικά με την TTIP, όμως είναι μια Καλή συνέχεια. Επίσης μας είπατε τη κατάσταση που επικρατεί ανάμεσα στην ε, κυβέρνηση των ΗΠΑ και στο Κογκρέσο. Πράγματι είναι προβληματικό αυτό που ακούσαμε. Όμως δεν έχουν όλοι τους ίδιους προβληματισμούς και τις ίδιες ανησυχίες στις ΗΠΑ σχετικά με την συμφωνία TTIP. Διαβάζοντας τι γίνεται στα κοινωνικά μέσα, έχω δει πολλές διαφορετικές ε, απόψεις και πολλή σύγχυση. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται διευκρίνηση του τι διακυβεύεται και τι όχι. Καλύτερη ενημέρωση λοιπόν. Χρειάζεται η συμφωνία αυτή να οδηγήσει σε πρόοδο. Και πιστεύω πως πρέπει να δείξουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως είμαστε διατεθειμένοι να αφιερωθούμε στην ε, συμφωνία TTIP και στο πώς αυτή θα δώσει τα μεγαλύτερα ωφέλη στους πολίτες της. Επίσης, όπως είπατε και εσείς, πιστεύω και εγώ να έχουμε θετικά αποτελέσματα και θα χαρώ πολύ να συζητήσω με τους υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές για να δούμε πώς θα καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε και να, και να ξεχωρίσουμε αυτές τις τόσο πολλές τροπολογίες και να δώσουμε λοιπόν στην, ε, με τη δική μας συνεισφορά στη συμφωνία TTIP την, ε, τα καλύτερα εφόδια για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών της. Πρέπει να γίνουν αλλαγές, αλλά εμείς πρέπει να φροντίσουμε οι αλλαγές αυτές να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα εστιάσω και εγώ, όπως και η Μαρίτια, σε ορισμένες τροπολογίες τις οποίες υποβάλαμε ως ε, πολιτική ομάδα. Καταρχάς να πω πως πιστεύω ότι ο αριθμός των τροπολογιών που έχουν συγκεντρωθεί δείχνει την νέα αντιμετώπιση αυτής της Επιτροπής και αυτού του Κοινοβουλίου την νέα αντιμετώπιση του ρόλου μας από αυτήν εδώ την Επιτροπή και από, αυτή, από το, εδώ το Κοινοβούλιο. Κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων διαπίστωσα, ε, διατύπωσα τη δική μου θέση και θα την επαναλάβω και τώρα. Χρειάζεται να δούμε τα ανοιχτά ερωτήματα σε αυτήν την συμφωνία και το πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να τα απαντήσει πρώτου προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, προτού, όπως είπε και η Μαρίτια, συνεχίσουμε και προτού λάβουμε την τελική μας θέση. Επίσης, θα ήθελα να σταθώ και σε αυτές τις πολλές ε, αντιφάσεις και στις πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις που έχουμε παρατηρήσει βλέπουμε πως αυτές οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν διαφορετικές ε, προτεραιότητες σίγουρα και πρέπει να δούμε τις επιμέρους λεπτομέρειες. Τρίτον, εμείς έχουμε αρκετά επικριτική άποψη και στάση σε αυτήν την συμφωνία και αυτό είναι γνωστό κιόλας. Διότι έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές αγορές. Με την ευρωπαϊκή αγορά που έχει και το ευρωπαϊκό και από πίσω της και με την αμερικανική αγορά. Και υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε αυτές τις δύο αγορές. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή και έχουμε υποβάλει σχετικές ε, τροπολογίες. Επίσης επικεντρωθήκαμε στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, στον τομέα των ε, δημόσιων υπηρεσιών, των ε, δημόσιων συμβάσεων, των υπηρεσιών κοινή ωφέλεια. Προσπαθήσαμε λοιπόν να επιστήσουμε την προσοχή σε θέματα που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά σε μια εμπορική συμφωνία, ναι. ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη. Και όπως ε, φάνηκε και από τις ε, τοποθετήσεις μας νωρίτερα με τον ε, Αντιπρόεδρο Κατάινεν, έχουμε διαφορετικές θέσεις για πολλά πράγματα με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αλλά φυσικά πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια κοινή θέση έτσι ώστε να ενισχύσουμε το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Τέλος, πιστεύω πως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε μια κοινή επικοινωνιακή στρατηγική. Και να δούμε ποια είναι η δική μας ευθύνη ως Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. διότι ακριβώς αυτές οι 898 τροπολογίες ε, το καθιστούν σαφές και εκτός από αυτές έχουμε και τις 14 γνωμοδοτήσεις που αναφέρατε. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να αποκρισταλώσουμε τις θέσεις όλων αυτών και να τις ε, ενώσουμε σε ένα περιεκτικό σχέδιο έκθεση. Ευχαριστώ. Κυρία Κέλλερ, το περιεχόμενο είναι γνωστό, αλλά η διαδικασία με ενδιαφέρει τώρα, είναι και αυτή σημαντική. Είναι πολύ σπουδαίο ως Επιτροπή Εμπορίου να χρησιμοποιήσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρογνωμοσύνη που έχουμε και τεχνογνωσία και από άλλες επιτροπές και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν όλες οι παράγραφοι και της επεξηγηματικής έκθεσης αναφέρουν τις πληροφορίες που θέλουμε να συγκεντρώσουμε και να συμπεριλάβουμε. Να μην το ξεχάσουμε αυτό επειδή είναι πολλές οι τροπολογίες. Αν λοιπόν ζητήσουμε από τις επιτροπές να πούν συγκεκριμένα ποιες θεωρούν τις σημαντικότερες παραγράφους και αυτό το κάνουν οι εισηγητές θα μπορέσουμε να μην περιοριστούμε σε συγκεκριμένους αριθμούς γιατί μερικές επιτροπές έχουν περισσότερες δικαιοδοσίες από άλλες. Επίσης πολύ καλό θα ήταν νομίζω να επιτρέψουμε στους γνωμοδοτούντες εισηγητές, στους συντάκτες γνωμοδοτήσεων δηλαδή, να παίξουν και αυτοί κάποιο ρόλο γιατί θα είναι πιο εύκολα όλα αυτά. Έχουν προβλεφθεί δύο τέτοιες συνεννοήσεις, θα έπρεπε ίσως να οργανωθεί και μία τρίτη. Γιατί γνωρίζετε ότι οι κατάλογοι ψηφοφορίας οδηγούν σε αντιμαχόμενες απόψεις κλπ. Και θα χρειαστεί χρόνος για να τα συζητηθούν και αυτά. Επίσης καλό θα ήταν νομίζω αν ήδη από την αρχή έχουμε τη δυνατότητα να γίνουν εναλλακτικές συμβιβαστικές προτάσεις γιατί το να συνδυαστούν τροπολογίες πολλών διαφορετικών κατευθύνσεων σε μία και μόνο συμβιβαστική δεν είναι πάντα εύκολο. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα λοιπόν να γίνει συμβιβασμός και επί ορισμένων συμβιβασμών. Συμβιβασμός του συμβιβασμού δηλαδή. Έτσι ώστε να γίνει η προσπάθεια μείωσης των, του αριθμού των ψηφοφοριών χωρίς να μειωθεί η σημασία τους. Επίσης ο εισηγητής θα μπορούσε να μας πει ποιες τροπολογίες καλύπτονται από συμβιβαστικές και ποιες όχι και ποιες θεωρεί σημαντικές να ψηφιστούν εκτός και συμβιβασμών. Θα ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν να ακολουθήσουμε μια τέτοια διαδικασία ώστε όλοι να γνωρίζουν τι ψηφίζουμε και μέχρι το τέλος Μαΐου βέβαια δεν είναι πολύ ο χρόνος αλλά θα παραμένουν μόνο 10 μέρες ας πούμε μέχρι την Ολομέλεια αφού ψηφίσουμε εμείς. Και επειδή θα κατατεθούν μάλλον τροπολογίες και στην Ολομέλεια δεν ξέρω ποιο είναι το καταλληλότερο χρονοδιάγραμμα. Πάντως ο στόχος πρέπει να είναι να φτάσουμε στην ψηφοφορία έχοντας όσο το δυνατόν πιο χρήσιμες πληροφορίες. Αυτά ήθελα να πω ε, διαδικαστικά. Begin. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και για την εκθεσή σας. Ε, με εξέπληξε θετικά. Με την ε, πρόταση κειμένου σας. Εγώ θα ήθελα απλώ να επαναλάβω τη θέση μας ε, για τη συμφωνία αυτή. Εμείς από το κίνημα 5 Αστέρια δεν θέλουμε την TTIP και γιατί, γιατί η συμφωνία αυτή δεν θα υποστηρίξει την επανεκβιομηχάνηση της Ευρώπης, ίσα ίσα θα την επιδονώσει, θα ε, αυξάνονται οι τιμές στην Ευρώπη, θα μειώνονται στην Αμερική και θα πιέσουν ε, έξω από τις αγορές τις επιχειρήσεις μας και θα βελτιώνουν τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Το διατρανωτικό εμπόριο θα πέσει κατά 40%, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θα έχουν ανταγωνισμό από πολύ μεγαλύτερους ε, ομίλους ε, και θα χάσουν πολύ σημαντικά πολύτιμα μερίδια αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην καλύτερη περίπτωση θα χαθούν 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέσω της συμφωνίας TIP και δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσουμε να ξαναπορροφήσουμε αυτές τις θέσεις εργασίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε ε, κάποια στοιχεία και κάποιες ε, τιμές οι οποίες δεν είναι ρεαλιστικές όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και ενώ θα έπρεπε να έχει προστατεύσει τους Ευρωπαίους πολίτες, τάσεται εναντίον τους. Επίσης ε, θα χαθεί και η κυριαρχία των κρατών μελών με αυθαίρετα δικαστήρια διατησίας και θα χαθούν τα προϊόντα ποιότητας και η TTIP θα έχει επενδύσει σε έρευνα και ανάπτυξη στις Ηνωμένε Πολιτείες που είναι χαμηλότερο το κόστος και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθεί στην ε, ε, τελευταία γραμμή. Υπάρχουν ε, κάποιες περιπτώσεις οι οποίες ήδη έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία βρίσκονται στα χέρια των λόμπι και των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς δεν είμαστε κατά το εμπορίου, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς όταν χρησιμοποιείται το εμπόριο για να δώσουμε τα προϊόντα μας σε αυτόν που θα κάνει τη μεγαλύτερη προσφορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και η συγκήτρια της Επιτροπής ΙΝΚΟ, ε, της νομοδότησης της ΙΝΚΟ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω τη θέση μου. Σας την έχω στείλει, την έχω πει και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Είμαι αναπληρώτρια εδώ στην Επιτροπή, οπότε την έχω πει και εδώ στην Επιτροπή. Θα ήθελα να κάνω τρεις-τέσσερις σύντομες παρατηρήσεις. Καταρχάς, θεωρώ ότι κατά την κατάρτιση της τελικής γνωμοδότησης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις. Πρώτον, τις δεσμεύσεις οι οποίες αναλήφθησαν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις ΗΠΑ για τις δημόσιες ε, υπηρεσίες κοινή ωφελίας, ε, κάτι το οποίο νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να γράψουμε κάτι λογικό για το κεφάλαιο των υπηρεσιών και νομίζω ότι και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη λεγόμενη υβριδική προσέγγιση. Δεύτερον, η Επίτροπος Μάλστρομ την περασμένο μήνα έκανε μια νέα πρόταση για το σύστημα επίλυσης διαφορών ε, ε, κράτους επενδυτή και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το περιλάβουμε στην τελική μας έκθεση. Θα ήταν ατυχές εάν το τελικό κείμενο δεν ε, περιλαμβάνει και την πρόταση της ε, Επιτρόπου. Μια τελευταία παρατήρηση για τον όλο τόνο της έκθεσης. Ε, πολύ καλή η εισαγωγική σας παρέμβαση, η οποία ήταν σε θετικό πνεύμα και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να μεταφραστεί και στο κείμενο. Αναφερθήκατε στις φιλοδοξίες ε, για την άλλη μεριά του Ατλαντικού, αλλά νομίζω ότι το αυτό ισχύει και για μας και για τη δική μας την έκθεση και θεωρώ ότι η έκθεση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποστείλει το μήνυμα ότι είμαστε κατά της συμφωνίας χωρίς να δούμε την ε, συμφωνία. Ε, Βασίζομαι λοιπόν στα αυτά που είπατε, ότι θα πρέπει να έχουμε ένα φιλόδοξο ε, κείμενο με θετικό πνεύμα. Κάτι τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, ως προς τη διαδικασία, όπως είπε και η προλαλήσασα, θεωρώ ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη και τα αποτελέσματα που έχουμε στις διάφορες επιτροπές, διότι εμείς ως Επιτροπή ΙΜΚΟ, για παράδειγμα, επενδύσαμε ενέργεια όχι μόνο στην κατάρτιση της γνωμοδότησης, αλλά επίσης ε, ε, οργανώθηκαν και αρκετές συνεδριάσεις και ακροάσεις επί του ζητήματος. Επομένως, θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την εμπειρογνωμοσύνη των διαφόρων επιτροπών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ντεβιτ Μάρτιν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Φυσικά, ε, πολύ καλή και πλήρης η έκθεσή σας. Ως προς τη διαδικασία, σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να προτείνουμε ε, πώς να διαχειριστείτε το θέμα αυτό. Νομίζω ότι ε, είστε ε, πλέον αρμόδιος να έχουμε μια καλή λύση. Εγώ δεν συμφωνώ όμως επειδή υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση να μην υπάρξει καμία περαιτέρω καθυστέρηση. Θα ήταν απαράδεκτο να περάσουμε πέρα από το ε, καλοκαίρι. Ε, θα πρέπει τον Ιούνιο να έχει εκφραστεί άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια και μάλιστα σαφέστατα. Πέντε τομείς μόνο. Ναι. Έχω και άλλους βέβαια αλλά πέντε θα ήθελα να θίξω. Ε, που θα θέλαμε να ενισχύσουμε να έχουμε μια κάποια διαφορετική απόχρωση στην έκθεση. Το πρώτο αφορά τα εργασιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα. Όπως είπαν ε, και διάφοροι άλλοι, ε, η TTIP μπορεί να έχει υψηλά επιχειρηματικά πρότυπα, αλλά θα πρέπει να έχει και στόχο ε, υψηλά εργασιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και κυρίως όλες οι συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας θα πρέπει να τηρηθούν βάσει της TTIP. Έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες για τις υπηρεσίες κοινή ωφελία και την εξαίρεση αυτών των υπηρεσιών. Η δήλωση της κυρίας ε, Μάλστρομ είναι αρκετά σαφής. Ε, δεν ξέρω αν είναι αρκετά σαφής ώστε να αναφέρεται στο κείμενο. Η σαφής μας όμως πρόθεση είναι να αποκλειστούν οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας και να μην περιλαμβάνονται στην TTIP. Και οι υπηρεσίες, ε, για παράδειγμα, υδάτων, η παιδεία, όλα αυτά θα πρέπει να βρίσκονται εκτός εντολής TTIP. Όσον αφορά το Συμβούλιο αυτό συνεργασίας, ε, εμείς ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διαδικασίες σε εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κυρίως για περιβαλλοντικές και κοινωνικές πολιτικές. Δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία απειλή για όλες αυτές τις πολιτικές λόγω της TTIP. Ε, η κόκκινη γραμμή για την ομάδα μου ε, δεν είναι η προστασία των επενδυτών αυτή καθεαυτή, αλλά το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα να νομοθετούμε. Οποιασδήποτε επενδυτική συμφωνία η οποία θα περιορίζει το δικαίωμα του νομοθετή για μας ε, είναι απαράδεκτη. Και επειδή προασπιζόμαστε τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η TTIP είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε η πολιτική μου ομάδα θεωρεί ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στην όλη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και θα πρέπει να έχουν και το δικαίωμα να κυρώσουν την TTIP όπως επίσης να την κυρώσουμε και εμείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι είναι τέτοια κλίμακα σε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν και τα εθνικά κοινοβούλια στη διαδικασία. Σε γενικέ γραμμέ, όπω σα είπα, θεωρούμε ευπρόσδεκτη την εκθεσή μα, διότι πηγαίνει προ την κατεύθυνση που θα θέλαμε να πηγαίνει και η Τίτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Τζούν. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω αυτά που είπε ο Ντέιβιντ και είμαι ανακουφισμένη που δεν θα ψηφίσουμε στις 7 Μαΐου γιατί έχουμε πιο σημαντική ψηφοφορία εκείνη τη μέρα για την επόμενη κυβέρνησή μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με ανακούφισε λοιπόν η αναβολή. Ο αριθμός των τροπολογιών δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και εκτός του Κοινοβουλίου για το TTIP. The of um, where there Και φυσικά θα είναι πολύ ενδιαφέρον φαντάζομαι εσείς και οι σκιώδεις να εξετάσετε πού μπορεί να υπάρξει κοινό έδαφος συμβιβασμών. Και για το Κοινοβούλιο θα φανεί ο ρόλος του στην διαπραγμάτευση για το TTIP και η κυρία Μάμστρομ μας είπε ποιο είναι το σχέδιο για το μέλλον. Είναι σημαντικό λοιπόν να καθορίσουμε πώς βλέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορισμένα θέματα. Οτιδήποτε στις τροπολογίες ζητάει να τεθούν σταθερά πρότυπα gold standards είναι σημαντικό. Πολλές τροπολογίες έλεγαν κάτι τέτοιο. Τώρα για τις δημόσιες υπηρεσίες, ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι είναι ζωτικό να έχουμε διατύπωση όπως εκείνη που λέει στην τροπολογία 397 δηλαδή όπου γίνεται λόγος για μείωση από την TTIP των υπηρεσιών κοινή ωφελία και κοινή οικονομικής ωφελία ή ενδιαφέροντος ή συμφέροντος είναι διότι πήραμε πληροφόρηση από νομικές υπηρεσίες και από εργαζόμενους που δείχνει ότι υπάρχουσες διατάξεις για αυτό το θέμα είναι πολύ αδύναμες και πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε την πολιτική θέληση να μην αποκλειστούν και οι δημόσιες υπηρεσίες. Να μπει αυτό στο σώμα το ίδιο του εγγράφου ότι οι δημόσιες υπηρεσίες μας δεν θα καλύπτονται από αυτή τη συμφωνία δεν περικόπτονται δηλαδή. Και τέλος για το ISDS. Δεν έχω ακόμη πιστεί καθόλου ότι υπάρχει λόγος να έχουμε συμφωνία ISDS με τη ΣΥΠΑ. Ένα όριμο νομικό σύστημα είναι απολύτως αρκετό για να μην χρειαστεί τέτοια συμφωνία. Αν ως Επιτροπή ΙΝΤΑ σκεφτούμε τι συζήτηση γίνεται μεταξύ επιτροπών θα δούμε ότι σημαντικότερη έγινε στην Ήτρε όπου εκλήθησαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κρίνουν το TTIP και στην ακρόαση εκείνη λοιπόν ακούστηκε η έκκληση των ΜΜΕ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ότι υφίστανται αθέμητο ανταγωνισμό από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι λοιπόν ζωτικό να βρεθεί κοινό τόπος και για αυτόν τον τομέα. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία για να φτάσουμε στην Ολομέλεια του Ιούνιο. Στούμε Βίμνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Διάβασα με μεγάλη προσοχή τις τροπολογίες και τις γνωμοδοτήσεις. ότι θέλουμε δηλαδή ψηλότερα πρότυπα για το περιβάλλον, για τα δικαιώματα των πολιτών, για την τροφιμική ασφάλεια, τα χημικά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρότυπα που να αναγνωριστούν και για την προστασία, την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών κλπ. Επίσης, και κατάλογος των θεμάτων που δεν θέλουμε να καλύπτει η συμφωνία. Οι άλλες επιτροπές βλέπουν κίνδυνο στη σύναψη συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ. Και υπάρχει όλο και μεγαλύτερη υποστήριξη για την διατήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων. Εγώ θα ήθελα η Κομισιόν να μας κάνει μια αξιολόγηση της συνθήκης TTIP στην τροπολογία 1 ας πούμε Ο συντάκτης από την ΚΟΕ μας λέει ότι το 0,5% που προβλεπόταν για τα 10 έτη προκύπτει απλώς από την κατάργηση των εσωτερικών τελειωνιακών φραγμών. Και ο καθηγητής Γκάμπριελ Μάγερ επίσης είπε το ίδιο. Θα ήθελα λοιπόν και εσείς να μου πείτε τι κερδίζουμε από το TTIP. Εγώ πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί έτσι μια τεράστια διατλαντική αγορά με πολλή γραφειοκρατία και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Και πιστεύω επίσης ότι όλο και περισσότερα εμπορεύματα θα διακινούνται με όλο και αρνητικότερες συνέπειες στο περιβάλλον, για το περιβάλλον. Πώς θα σεβαστούμε τους κλιματολογικούς μας στόχους. Πρέπει το εμπόριο να μην ασκείται εις βάρος των τρίτων χωρών. Και εγώ νομίζω ότι εδώ πρόκειται για το πρόγραμμα του Business Europe ως έχει, χωρίς αλλαγή. Ανησυχεί ο κόσμος για το TTIP. Να, εδώ μοίρασα αυτά τα πράγματα με ένα ε, Ολλανδικό λογοπαίγνιο επάνω που λέει TTIP is not my cup of tea. Κύριε σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι το πρώτο πρέπει να, που πρέπει να αναρωτηθούμε όταν βλέπουμε αυτόν τον τεράστιο όγκο τροπολογιών είναι τι, τι θα τις κάνουμε και τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτές τις τροπολογίες. Και πιστεύω πως πρέπει να κάνουμε μια επιλογή σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την έκθεση και το ποιο ρόλο θέλουμε να παίξει σε αυτή τη διαδικασία. Θα θεωρήσουμε δηλαδή αυτή την έκθεση σαν συνέχεια εκείνης που κάναμε πριν από δύο χρόνια, ως φυσική συνέχεια λοιπόν εκείνης της ε, έκθεσης. Θα τη δούμε ως ε, μια έκθεση που παρακολουθεί τις ε, τρέχουσες διαπραγματεύσεις και θα ελέγχει κατά πόσο οι διαπραγματεύσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν αυτά που είχαμε γράψει στην προηγούμενη έκθεση ή η άλλη προσέγγιση να κάνουμε ένα νέο ψήφισμα το οποίο θα αντικαταστήσει το παλαιότερο ψήφισμα και κατά μια νέα εντολή για ένα νέο κοινοβούλιο. Διότι πιστεύω πως ε, αυτές είναι οι δύο επιλογές και δεν μπορούμε να τις συνδυάσουμε. Κάποιες τροπολογίες ε, είναι προς αυτή τη μία κατεύθυνση και κάποιες προς την άλλη. Εγώ είμαι υπέρ της πρώτης λύσης και της πρώτης επιλογής και δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι αφού δεν μπόρεσαν να περάσουν οι δικές μου τροπολογίες την προηγούμενη φορά, ε, να περάσουν τώρα. Δεν πιστεύω πως αυτό είναι σωστό. Και πιστεύω πως επίσης δεν είναι σωστό να μεταφέρουμε το τέρμα σε άλλο σημείο του γηπέδου, όπως γίνεται τώρα με τις διαπραγματεύσεις σε σχέση με τις παλαιότερες, διότι διακυβεύεται η αξιοπιστία μας όντως ένας ε, σοβαρός εταίρος που προσπαθεί να προωθήσει μια εμπορική συμφωνία. Εάν επιλέξουμε τη δική μου γραμμή, δηλαδή να χτίσουμε πάνω σε αυτό που έχουμε, τότε δεν θα δημιουργήσουμε νέες κόκκινες γραμμές, δεν θα πούμε «Α, και ξέρετε, ξεχάσαμε και αυτό, ναι, πάρτε το τώρα». Όχι. Θα χτίσουμε λοιπόν πάνω σε αυτά που έχουμε και πιστεύω πως υπάρχει η ανάγκη να το κάνουμε, πως έχουμε τη δυνατότητα μέσω των πολύ καλών προτάσεων που έχω διαβάσει να το πράξουμε και πολλές από τις τροπολογίες κάνουν ακριβώς ε, αυτό. Για παράδειγμα, ζητούν απελευθέρωση στις ε, θεωρήσεις. Βλέπω ότι πολλοί συνάδελφοι το έχουν ζητήσει. Ε, μιλούν για τις υπηρεσίες ε, μεταφορών, για τους δασμούς, για τα μη δασμολογικά εμπόδια. Όπως και στην έκθεση Μορέιρα, έτσι και σε αυτή πιστεύω πως πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτούς τους τομείς. Από την άλλη, πολλές από τις εγνωμοδοτήσεις που έχω διαβάσει και να πω εδώ ότι φυσικά και πρέπει να τις σεβαστούμε αλλά να μην ξεχνάμε και το δικό μας ρόλο ως αρμόδια επιτροπή έχω δει λοιπόν πάρα πολλές νέες κόκκινες γραμμές και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να μην δημιουργήσουμε νέες κόκκινες γραμμές που θα αλλάξουν την κατεύθυνση που έχουμε μέχρι τώρα. Υπάρχουν λοιπόν πολλές εγνωμοδοτήσεις που λένε το αντελώς αντίθετο από όσα ξέρουμε μέχρι τώρα. Χρειάζεται λοιπόν ε, να αναρωτηθούμε και να δούμε εάν οι γνωμοδοτήσει των επιτροπών δημιουργούν νέες κόκκινες γραμμές. Έπειτα, το θέμα του ISDS. Πιστεύω πως έχουν γίνει τόσες πολλές συζητήσεις για την επιλύστη φορών επενδυτή και κράτους που δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε περαιτέρω αυτή τη στιγμή. Με χαρά μου όμως θα ακούσω την δική σας πρόταση για τη διατύπωση, συνάδελφε από τους σοσιαλδημοκράτες, ότι δηλαδή δεν είστε ακριβώς αντίθετος με αυτή τη συμφωνία, αλλά αν υπάρξει αυτή η συμφωνία πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα όλων κτλ. Βέβαια, αυτή η έκφραση που βλέπω εδώ, το, τα ρυθμιστικά δικαιώματα, πρέπει να δούμε και τι σημαίνουν και να δούμε τι σημαίνει το να μην απειλούνται τα ρυθμιστικά δικαιώματα. Μπορεί δηλαδή να έχει το δικαίωμα να κάνει κάποια πράγματα τα οποία όμως θα έχουν και ένα κόστος από πλευρά του κράτους. Χρειάζονται λοιπόν καλές διατάξεις σχετικά με το ISDS για την ε, προστασία των επενδυτών και οι καλές αυτές διατάξεις θα βοηθήσουν τον νομοθέτη να δει τις συνέπειες των διακρίσεων αυτών ή των ε, άλλων πράξεων ή των απαλωτριώσεων χωρίς αποζημίωση, για παράδειγμα. Και πιστεύω πως ε, συμμεριζόμαστε όλη αυτή την άποψη, το εύχομαι τουλάχιστον, διότι έτσι με μια καλή διατύπωση θα καταφέρουμε να έχουμε ε, μια επικοδομητική βάση για το μέλλον. Ο κύριος Προύστ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ναι. ναι, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί πολλά έχουν υποθεί από άλλους. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τον μεγάλο αριθμό των τροπολογιών. εφόσον είναι επικοδομητικές και παιδαγωγικές στο χαρακτήρα τους. Και εγώ θέλησα να καταθέσω τροπολογίες για να είμαστε πιο σαφείς Όλοι περιμένουν αυτό, σαφήνεια και δέσμευση των κοινοβουλευτικών για αυτό το σημαντικό θέμα. Όχι για να αντιταχθούμε συστηματικά, αλλά με συγκεκριμένες προτάσεις που θα δώσουν μια δεύτερη εντολή διαπραγματεύσεων για να είμαστε συγκεκριμενότεροι. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον πρόεδρο και τους εισηγητές για να τηρήσουν αυτήν την γραμμή επικοδομητική και παιδαγωγική. Ίσως δεν Χριστόφορε γιατί μίλησε και για το ISDS. Το παράδειγμα σχέσεων της εταιρείας Σουέζ με την Αργεντινή ίσως να μας δείχνει προς τα που κινούμεθα για τη μελλοντική ISDS που ίσως να αλλάξει και όνομα και να προστατεύει και τα κράτη και τους επενδυτάς και επενδύτριες. Ωραία, ευχαριστούμε. Ο Ιγνάτιος από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Είναι σαφές ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, το συγκεκριμένο ψήφισμα είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Θα πρέπει σαφώς ε, να υπάρξει ένα σαφές μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς υποστήριξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας ε, TTIP. Είναι σαφές ότι το ψήφισμα θα εγκριθεί σε μια πολύ σημαντική και δύσκολη χρονική συγκυρία στις διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΠ, επομένως ε, θα έχει σημαντική επιρροή. Αναφερθήκατε στις συζητήσεις ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να είμαστε σε αναμονή. Από τα μηνύματα που λαμβάνουμε, η νομοθεσία ε, TPA μπορεί να περάσει σύντομα από το Κογκρέσο, αλλά σίγουρα δεν θα είναι μια απλή συζήτηση και επομένως πρέπει να παρακολουθούμε στενά τι ακριβώς περιλαμβάνεται σε αυτή τη συμφων... στην νομοθεσία TPA, η οποία θα συζητηθεί στο Κογκρέσο, ώστε να αποφύγουμε και μηνύματα από πλευράς Κογκρέσου, ε, τα οποία θα δυσκολέψουν τις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι εμπιστευόμαστε ιδιαίτερα και εσά κύριε Πρόεδρε και τα μέλη της Επιτροπής σας ε, για να μας οδηγήσετε σε ένα ψήφισμα το οποίο θα βοηθήσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης ε, επισημάνατε ποιοι είναι οι πέντε τομεί που είναι οι πιο δύσκολοι και είμαι βέβαιος ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε προκειμένου να εξευρεθούν συμβιβασμοί οι οποίοι θα τύχουν ευρεία υποστήριξη. Νομίζω ότι και η Επιτροπή σας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ε, το στηρίξει αυτό. Δεν θα σχολιάσω καθόλου την ισουία. Δύο σχόλια να κάνω. Για το θέμα της προστασίας των επενδυτών και τη διατησία σε θέματα ε, επενδύσεων θεωρούμε ότι ε, η σωστή άγουσα είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος και η Επίτροπο Μάλστρο θα επανέλθει στην Επιτροπή σας στις 7 Μαΐου με πολύ συγκεκριμένες υποδείξεις για το τι ακριβώς ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να προωθήσουμε ε, σε πλαίσια μεταρρύθμισης ενός συστήματος προστασίας των επενδυτών και της διαδιαιτησίας. Όσον αφορά των υπηρεσιο... τις υπηρεσίες. Νομίζω ότι κάποιοι από εσάς αναφερθήκατε στην κοινή δήλωση Επιτρόπου Μάλστρομ και του πρέσβη Φρόμαντ και επίσης θα ήθελα να επιστήσω και την προσοχή σας και στην τρίτη παράγραφο της συγκεκριμένη δήλωσης διότι νομίζω ότι εκεί ε, περιλαμβάνονται σαφέστατα μηνύματα. Καμία δέσμευση για απελευθέρωση δημοσίων υπηρεσιών, δεν υπάρχει κανένα πρόσκομα ε, για ε, συγκεκριμένες υπηρεσίες οι οποίες ε, παρέχονται από το δημόσιο τομέα και κανένα πρόσκομα στο να επανέλθουν στο δημόσιο τομέα υπηρεσίες οι οποίες στο παρελθόν αποτελούσαν αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι σαφέστερο το μήνυμα για τις δημόσιες υπηρεσίες. Ε, τέλος, δύο λόγια όσον αφορά το θέμα της βιωσιμότητας. Ε, είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό θα είναι ένα από τα πολύ σημαντικά κεφάλαια της συγκεκριμένη συμφωνίας. Στόχος μας είναι να ε, έχουμε έτοιμα στις προτάσεις μας πριν από το γύρο διαπραγματεύσεων του Ιουλίου και αυτό το οποίο θεωρούμε είναι να υπάρξει μια συμφωνία για τα θέματα αυτά η οποία θα υπερβαίνει τα όσα έχουν κάνει μέχρι τούδε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες στις άλλες του συμφωνίες. Αυτά λοιπόν ε, εν είδη σύντομων σχολείων και όπως σας είπα προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας και με την Επιτροπή σας διότι περνάμε σε μια πολύ σημαντική φάση των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους. Θα ήθελα τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, να μου επιτρέψετε να κάνω ορισμένε παρατηρήσει και ορισμένα σχόλια πριν το τέλο. Πράγματι, όπω ε, φάνηκε και από αυτήν την ε, σύντομη συζήτηση, έχουμε καταφέρει να, εντοπίσει, να εντοπίσουμε ορισμένου ε, τομεί που θεωρούμε δύσκολου ή αμφιλεγόμενου. Εκτός λοιπόν από αυτούς τους τομείς, Πιστεύω πως όλες οι τροπολογίες και οι γνωμοδοτήσεις που έχω στη διάθεση μέχρι στιγμής πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση, προς μια βελτίωση δηλαδή των λεπτομεριών της συμφωνίας αυτής. Και αυτή είναι και η συνεισφορά αυτής της έκθεσης. Πιστεύω πως είναι προς το δικό μας συμφέρον να αναλάβουμε δράση απέναντι στην ε, συμφωνία TTIP έτσι ώστε να δώσουμε μία αποφασιστική στάση στην, για την ε, συμφωνία αυτή. Πιστεύω πως ε, έτσι θα καταφέρουμε να οδηγηθούμε σε καλά αποτελέσματα. Τώρα, φάνηκε ξεκάθαρα πως το ISTS είναι ο πιο αμφιλεγόμενος τομέας και ο Κινάσιο είναι ο αρμόδιος και έχει έρθει στην Επιτροπή μας, μας έχει παρουσιάσει πάρα πολλές ε, φορές την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Θα πάει και στο Συμβούλιο για να παρουσιάσει εκεί το νέο μοντέλο εργασίας και επειδή προβλέπεται η συμμεταχείριση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου αναμένω να έρχεται όχι μόνο ο αγαπητός Ιγνάσιο, αλλά και η ίδια η Επίτροπος εδώ σε εμάς, στην Επιτροπή μας, έτσι ώστε να μπορέσει να συζητήσει μαζί μας. Και φυσικά τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων θα ενσωματωθούν στην έκθεσή μας, σίγουρα. Τώρα, όσον αφορά τις ε, δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες κοινή ωφέλεια, ε, φυσικά αναγνωρίζω πω πρόκειται για ένα πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, διότι κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικές ε, συνθήκες και διαφορετική αντιμετώπιση. Πιστεύω όμως ότι ένα άνοιγμα του τομέα αυτού πρέπει να συμβεί μόνο εφόσον εμείς και δηλαδή οι τοπικές αρχές το επιθυμούν και εδώ έχει και η Μαρή ο Ιγνάσιο δίκιο όταν τοποθετήθηκαν ε, για αυτή την ε, δήλωση μάλιστα Πρέπει δηλαδή να γίνει, είναι καλό να γίνει, αλλά υπό προϋποθέσεις και εφόσον υπάρχει αυτή η επιθυμία. Χρειάζεται όμως να ε, εξετάσουμε τις λεπτομέρειες ξανά, διότι υπάρχουν οι υπηρεσίες, κοινές υπηρεσίες, ε, δημόσιες υπηρεσίες κοινή ωφέλεια, οι οποίες δεν επιχορηγούνται από το κράτος, προστατεύονται όμως τρόπον την από αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί στην επιλογή της διατύπωσης. Επίσης, το θέμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Είναι για μένα κεντρικό κομβικό σημείο, διότι συμπεριλαμβάνει πάρα πολλές ε, περιπτώσεις ε, κινδύνων. Φυσικά, αθέμητος ανταγωνισμός, η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ε, προϊόντων και των παροχών υπηρεσιών, αλλά και υπάρχει ο κίνδυνος του κοινωνικού ντάμπινγκ. Πρέπει να διατηρηθούν επίσης αυτά τα 8 πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε πως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως σας είπα και στην αρχή της συνεδρίασης, είχα πάει στο Βιετνάμ και είδα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για την TTP ζητούν από το Βιετνάμ να κυρώσει και να εφαρμόσει αυτά τα οχτώ πρότυπα του ε, Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Το οποίο θα τα καταστήσει φυσικά δεσμευτικά. Αυτό δηλαδή είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε από τη μία ζητούν από τους εταίρους τους στη συμφωνία TTP να δεσμευτούν για τα 8 πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, όμως στη δική μας περίπτωση στη συμφωνία TTIP δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται λοιπόν μία διευκρίνηση και χρειάζεται μία σαφή τοποθέτηση από τη μεριά τους. Επίσης, ρυθμιστική συνεργασία. Ο David Μάρτιν αναφέρθηκε σε αυτήν. Είναι πραγματικά κάτι καινούριο για πολλούς από εσάς. Δεν την συζητήσαμε όσο ε, θα έπρεπε ίσως ε, στα πλαίσια της έκθεσης ε, Βιτάλ Μορέιρα. αλλά πιστεύω πως δεν υπάρχει κάτι το αμφιλεγόμενο εδώ. Πιστεύω πως συγκλίνουν οι απόψεις μας, θέλουμε υψηλά πρότυπα. Όμως, υπάρχει το θέμα των ε, ρυθμίσεων και των πράξεων ε, κατά εξουσιοδότηση εκτελεστικών ε, πράξεων. Υπάρχει δηλαδή θέμα δομής το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Όμως βλέπω πως σε αυτό το θέμα οι περισσότερες τροπολογίες συγκλίνουν ή πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Έπειτα, να κάνω και έναν μικρό απολογισμό για το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και πώς προχωρούμε. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο από το να βασιστούμε απλά στην έκθεση Μοραΐρα και να συγκεντρώσουμε απλά γεγονότα. Χρειάζεται περισσότερη λεπτομερής αναφορά και μια ευρύτερη συζήτηση και μια πιο δημόσια συζήτηση με όλους τους εκπροσώπους και φυσικά και εκπροσώπους των ε, πολιτών, των ψηφοφόρων μας. για να δούμε τι σε προτάσεις ενδεχομένως προκύψουν. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε τον απολογισμό μας και να αναλογιστούμε για τα όσα έχουμε κάνει και για να δούμε τι πρέπει να περιμένουμε από το μέλλον. Και τώρα ξαναφτάνω σε αυτές τις 898 τροπολογίες και στις 14 νομοδοτήσεις από τις υπόλοιπες επιτροπές. Να πω ότι όλα αυτά είναι προς δικό μας όφελος, διότι έχουμε γνωμοδοτήσεις που έχουν συνταχθεί από ομάδες εμπειρογνωμόνων και από την Επιτροπή Πολιτισμού και από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και από την Επιτροπή ΙΝΚΟ, ε, οι οποίες γνωμοδοτήσεις ασχολούνται με επιμέρους σημεία και μπαίνουν σε λεπτομέρειες, σε σημεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να εξετάσουμε τόσο ενδελεχώς. Θα εμπλουτίσουν λοιπόν τη δική μας ε, έκθεση και τη δική μας δουλειά. Ωστόσο πρέπει να προσπαθήσουμε να οδηγηθούμε και σε έναν συμβιβασμό με όλες αυτές τις διαφορετικές κατευθύνσεις που παίρνουν αυτές οι γνωμοδοτήσεις. Λοιπόν, μέσα στην επόμενη εβδομάδα περιμένω από εσάς να δείτε πώς θα βρούμε συμβιβασμούς έτσι ώστε να ενώσουμε τις ε, τροπολογίες, έτσι ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε μια έκθεση για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Πιστεύω πως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και οι 898 τροπολογίες σας μην σας τρομάζουν. Υπήρξαν άλλες σε περιπτώσεις όπου είχαμε 3.000 τροπολογίες. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι με την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει, με το συμβιβαστικό πνεύμα και το πνεύμα συνεργασίας θα καταφέρουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, μια αποφασισμένη και σταθερή θέση έτσι, λοιπόν, με όλα αυτά θα οδηγηθούμε σε μια επικοδομητική εργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Yes, uh, dear colleagues, this was a lot. κύριοι συνάδελφοι, αυτό ήταν δυστυχώς το τελευταίο θέμα σήμερα. Πρώτης ώρας του τελείωσε. Μισή ώρα νωρίτερα. Θα σας ξαναδούμε αύριο το πρωί στις 9. Χαίρετε.